Εντάξει, κάπω καθυστερημένο. Είναι μια κοινή συζήτηση για τον προπολογισμό το 2014 και το 2015. Έχουμε μια σειρά εκθέσεων και μιας και πρόκειται για κοινή συζήτηση. Η πρώτη έκθεση είναι της κυρίας Γκαρδία Ζαμπάλ Ρουμπιάλ και της κυρίας Χολμάιερ. Επτά είναι οι, οι εκθέσεις του κύριου Ντεπρέ και μετά κοινή έκθεση Ντεπρέ και Λεβαντόφσκι θα περάσουμε πάρα αυτά στη συζήτηση και δίνω το λόγο λοιπόν στους συζητητές για τέσσερα λεπτά. Η κυρία Γκαρτεζιαμπέλ, Ρούμπιερ, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ναι, η αλήθεια είναι σωρεύτηκε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών κάπως η δουλειά και γι' αυτό σήμερα έχουμε τόσες πολλές εκθέσεις που θα πρέπει να συζητήσουμε και αύριο να ψηφίσουμε. Η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με αυτά τα οποία καταλήξαμε ως συμφωνία για τον προϋπολογισμό 2015 ούτε και για τους αναγκαίους ε, διορθωτικούς προϋπολογισμούς ε, και αυτό χάρη στο έργο πολλών που ενεπλάξαν σε αυτή την προσπάθεια και που είναι σήμερα στην Ολομέλεια. Θα ήθελα να ξεκινήσω λοιπόν την παρέμβασή μου ευχαριστώντας την Επίτροπο Γεωργίευα και τους υπαλλήλους και την Ιταλική ε, Προεδρία και τον Ιταλό Πρέσβη και όλους τους συναδέλφους διότι συνεργαστήκαμε πάρα πολύ έντονα τους τελευταίους μήνες για να καταλήξουμε σε αυτή τη συμφωνία. Και έλεγα τίποτα δεν προανήγγειλε ότι θα είχαμε έγκαιρα μια συμφωνία διότι ήταν πολύ μακριά η μία θέση από την άλλη και παρεξέκλειναν οι θέσεις. Η αρχική θέση δηλαδή η πρόταση του Συμβουλίου και η θέση του ε, Κοινοβουλίου. Αλλά απέκλειναν οι θέσεις και σε σχέση με τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο των 28 κρατών μελών. Υπήρχαν αποκλίνουσες προτάσει, υπήρχαν επιφυλάξεις μεταξύ θεσμικών οργάνων, μεταξύ χωρών, αμφιβολίε για τα αριθμητικά μεγέθη και σε σχέση και με τα κονδύλια τα οποία θα έπρεπε να διατεθούν. Έχουμε λοιπόν τα τρία θέματα που έπρεπε να επιληθούν. Πώς θα ολοκληρωνόταν το 2014, πώς θα ξεκινούσαμε και θα αντιμετωπίζαμε το 2015 και ένα πρόγραμμα για να αντιμετωπιστούν οι συσσωρευτήσεις μη εκτελεστήσεις πληρωμές. Και ως εισηγήτρια πρέπει να πω ότι δεν είμαι ε, ούτε για τα αριθμητικά μεγέθη, ούτε για τη λειτουργία, ούτε για την απουσία του πολιτικού κιόλα περιεχομένου σε συζήτηση. Όμως ένα ολόκληρο χρόνο εργαστήκαμε για να καταλήξουμε σε αυτή τη συμφωνία να καταλήξουμε σε ένα προπολογισμό. Και ξέρω ότι η τελευταία πρόταση που είχαμε στο τραπέζι και που σήμερα είναι αναγκαίο να πούμε ότι πρέπει να υποστηρίξετε αύριο ψηφίζοντα ήταν η καλύτερη που μπορούσαμε να επιτύχουμε. Διότι 4 δις 600 εκατομμύρια επιπλέον δίνει αυτή η πρόταση σε σχέση με τα προγράμματα που πρέπει να εκτελεστούν. 4 δις 600 εκατομμύρια για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις για να μπορέσουν να συνεχίσουν με τις μεγαλύτερες ανάγκες το έργο τους και να υπάρξει το έργο αυτό για την οικονομική ανάκαμψη και για τους γεωργούς που με το βέτο της Ρωσίας για την εξαγωγή των προϊόντων τους επλήγησαν και για να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη τις ανάγκες των πολιτών γιατί περί αυτού πρόκειται σε αυτόν τον προϋπολογισμό για ένα ευρωπαϊκό προϋπολογισμό να λάβουμε υπόψη τις ανάγκες των πολιτών με υποτροφίες, με την βοήθεια βοήθεια όσον αφορά την, ε, τις υποδομές τους ε, πρόσφυγες από τη Μέση Ανατολή για την δημιουργία επίσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, τράπεζα επισητιστικών επίσης καταπολέμηση των ακροτηριασμών γενετής, γενετι, γεννητικών οργάνων των γυναικών δώσαμε μάχη για όλα αυτά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η εναλλακτική λύση έναντι όλων αυτών θα ήταν να μην υπάρχει συμφωνία να μην έχουμε προϋπολισμό για το 2015 να χάσουμε δώσουμε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα 4 δις 600 εκατομμύρια επιπλέον που δεν προβλεπόντουσαν στο προϋπολογισμό της Ένωσης. Θα διακυβευόταν λοιπόν το πρόγραμμα επενδύσεων που η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις μας παρουσίασε διότι βασίζεται 100% στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Ξέρουμε ότι αυτά τα 4 δις 600 εκατομμύρια δεν επαρκούν διότι το πρόβλημα των μη εκτελεστησών πληρωμών είναι μεγαλύτερο. Γι' αυτό τονίζουμε να αναζητηθεί συμφωνία, συμβιβασμό με το Συμβούλιο για να μπορέσουμε από την έναρξη του 2015 να έχουμε ένα αυθεντικό πρόγραμμα εργασίας για να χτυπηθεί το πρόβλημα στη ρίζα του. Διότι όσον αφορά το 1% των δαπανών ΑΕΠ δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Έχουμε ένα πρόβλημα εσόδων. Και όταν έχουμε περικοπή ή συστολή του προπολογισμού, η λύση είναι η αύξηση των ιδίων πόρων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μείωση δηλαδή των εθνικών συνεισφορών. Λυπούμε ότι με τι καθυστερήσει που υπάρχουν έχουν παγώσει τα πράγματα και δεν καταλήξαμε σε συμφωνία. Γι' αυτό πιστεύω ότι η ομάδα υψηλών αξιωματούχων για του ίδιου πόρου είναι απόλυτα αναγκαία. Περισσότερο αναγκαία από ό,τι στο παρελθόν παρελθόν για να υπάρξει ένας ισχυρός προϋπολογισμός που θα χρηματοδοτείται επαρκώς και σωστά και να μπορέσει πραγματικά να αντιμετωπίσει τις ανάγκες πέρα από λογιστικές ανάγκες. Αυτό χρειαζόμαστε στο μέλλον. Ευχαριστώ. Uh, and thank you. Σας ευχαριστώ και θα... Είμαι λίγο πιο επίκης προς τους συζητητές από ότι προς τους ομιλητές, αλλά σας παρακαλώ να τελειώ το χρόνο Η κυρία Χόλμα είναι η επόμενη ομιλητρία για τέσσερα λεπτά. Έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Επίτροπε, να να χαιρετήσω και την Προεδρία του Συμβουλίου. Θα ήθελα εξ αρχής να ευχαριστήσω να σας ευχαριστήσω γιατί θεωρώ ότι μετά από ένα μαραθώνιο διαπραγματεύσεων καταφέραμε τελικά ο, η πρόεδρος ε, της Επιτροπής και η συνάδελφος που υπερασπίζεται τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ε, αντιπροσωπεία, αγαπητέ Χωσέ Μαγγελ και τον κύριο Ντεπρέ βλέπω επίσης και όλοι καταφέραμε μετά από ένα μαραθώνιο διαπραγματεύσεων να περάσουμε ένα προπολογισμό όπου οι συντονιστές σε καμία περίπτωση δεν ήταν αρχικά σύμφωνοι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το Ηράκλειο αυτό έργο. Να ευχαριστήσω και την Επίτροπο κατά δεύτερον, η οποία με την δική της ομάδα πολέμησε για να περάσει ο προπολογισμό αυτός και μετά την Ιταλική Προεδρία όπου στην αρχή υπήρχαν μεγάλες δυσκολίες, αλλά εν πάση περιπτώσει στο τέλος όλοι συμφώνησαν και καταφέραν να πετύχουν το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Δεν είναι το βέλτιστο, αλλά τουλάχιστον είναι μία οδός, ένας δρόμος. Και επίσης ό,τι αφορά τα άλλα θεσμικά όργανα, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για τα διοικητικά έξοδα, τα οποία μας τα προέβαλαν με διαφανή τρόπο και το ΔΕΚ που τελικά καταφέραμε να συμφωνήσουμε για μία λύση για τους νέους δικαστές και για το θέμα το, του εμπορίου σε ό,τι αφορά τις δύο επιτροπές από πλευράς του δικαστηρίου και επίσης από πλευράς του Κοινοβουλίου για τη συνεργασία την οποία κάναμε σε ό,τι αφορά την συνεργασία μεταξύ οικονομικής ε, Επιτροπής και Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων. Στα άλλα θεσμικά όργανα, λοιπόν, τα προβλήματα δεν ήταν τόσο σημαντικά όπως ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μας ε, τυράνιζαν πραγματικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι παλιοί λογαριασμοί και θα ήθελα να πω το εξή. Δεν μπορούμε σε τελική ανάλυση με τον νέο προπολογισμό που έχουμε να πληρώνουμε μόνο παλιούς λογαριασμούς. Θα πρέπει τα προγράμματα τα οποία έχουμε και τα οποία επί σειρά επί ε, σειρά ετών ε, τα καταστήσαμε, να τα φρενάρουμε, να τα τρενάρουμε τεχνητά, προκειμένου να μπορέσουμε να εγγυηθούμε τις πληρωμές. Αυτή είναι μια πραγματικά απαράτακτη κατάσταση και γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι μεγάλη επιτυχία που τουλάχιστον το θέμα του σχεδίου των πληρωμών και των εγγυήσεων εκτέλεση του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου το συμπεριλάβαμε στη συζήτηση. Και θέλουμε να πετύχουμε μία λύση. Ελπίζω δε το Συμβούλιο και τα κρατημέλη να είναι πιο παρόντες σε αυτές τις συνεδριάσεις και το λέω ξεκάθαρα σε σχέση με την συνεδρίαση για τους ε, οργανισμούς, την ανάλυση των εργασιών τους και την σχετική χρηματοδότηση, πρικοδότησή τους. Καλό λοιπόν το Συμβούλιο εκ βάθους καρδίας να κοιτάξει το θέμα του σχεδίου ε, πληρωμών και των ε, νέων προγραμμάτων γιατί θέλουμε να τα πετύχουμε αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Κοινοβούλιο δεν έμεινε ξεροκέφαλα στα παραπάνω ποσά που ζητούσε αρχικά, αλλά κάτσαμε διαπραγματευτήκαμε μαζί σας, κάναμε και υποχωρήσεις, αλλά θέλουμε αντίστοιχα και εσάς και εσείς στην νόμιμη αξίωσή μας να πληρωθούν οι παλιοί λογαριασμοί προκειμένου να μην χρεώνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση διαρκώς να ανταποκριθείτε και να καταστεί και αυτό ο βασικό σας συμφέρον. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής είναι ο εισηγητής μας, ο κύριος Δεπρέ, ο οποίος θα μιλήσει για τέσσερα λεπτά, είναι αρμόδιος για επτά ε, εκθέσεις και μία εκθέση είναι αρμόδιος με τον κύριο Λεβαντόφσκι. Ε, κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, στην εκκίνηση των πραγματές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω της Επιτροπής Ορπολογισμών καθόρισε τρεις προτεραιότητες. Τρεις στόχους. Πρώτος στόχος, σταθεροποίηση και ή δυνατόν μείωση του ανησυχητικού επίπεδου των μη πληρωμένων λογαριασμών. 25 ε, δισεκατομμύρια το τέλος του 2014. Πρώτη προτεραιότητα λοιπόν ήταν σταθεροποίηση των απλήρωτων λογαριασμών. Δεύτερος στόχος, ε, να σταματήσει αντιπαράθεση με το Συμβούλιο όσον αφορά το καθεστώς των ειδικών μέσων, κυρίως για τις πληρωμές. Τρίτος στόχος, βασικός στόχος να συμφωνήσουμε με τα δύο άλλα θεσμικά οργάνα όσον αφορά την κατεπίγουσα εφαρμογή σχεδίου ε, πληρωμής ε, των ε, μη πληρωμένων λογαριασμών. Ποια είναι τα συμπεράσματα μπορούμε να συναγάγουμε μετά από τι πολλέ εβδομάδε διαπραγματεύσεων. Τέλο πάντων, δεν θα έλεγα διαπραγματεύσει, διότι περισσότερε συνεδριάσει βασίστηκαν στο να ακούμε το Συμβούλιο να λέει ότι δεν ήταν δυστυχώ σε θέση να έχει κοινή θέση. Τώρα, όσον αφορά τον απολογισμό, τις πιστώσεις πληρωμών καταρχάς. Η συμφωνία προβλέπει για το 2014 και μόνο συμπροματικά ανωπά χρήματα όπως λέγεται 3 δισεκατομμύρια 529 εκατομμύρια δηλαδή 2 τρίτα εκείνων που απαιτούσαμε στην αρχή και διευκρινίζω λέγοντας ότι είχαμε δεσμευτεί να ζητήσουμε εκείνο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρούσε ως απαραίτητο, δηλαδή 4,7 δις το 2014, ούτως ώστε η κατάσταση να μην συνεχίζει να επιδεινώνεται όσον αφορά τους απλήρωτους λογαριασμούς. Δεύτερον, όσον αφορά το δημοσιονομικό καθεστώς των ειδικών μέσων, διαφορά μεταξύ θέσεως του Συμβουλίου και της θέσεως του Ευρωκοινοβουλίου δεν μπόρεσε να καλυφθεί η διαφορά. Λύση ουδέτερη είναι στα 350 εκατομμύρια ε, στις πιστώσεις μη χρησιμοποιηθέντα θέματα. Όσον αφορά το σχέδιο καθάρισης που είναι σημαντικό των αυξανόμενου ποσού των απλήρωτων λογαριασμών είναι μια συμφωνία που μπόρεσε να επιτευχθεί. Θα πρέπει να παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Μάρτιο 2015 μια επίκαιρη αξιολόγηση του συνολικού ποσού των απληρώτων και να προτείνει εναλλακτικέ λύσει. Τα τέθεσμικά όργανα θα δεσμευτούν να εφαρμόσουν ένα σχέδιο στη φάση αυτή και ζητάμε να επισοποιήσει απέναντί μας τη δέσμευση ότι το, θα συμφωνηθεί το πρόγραμμα αυτό από τα τρία θεσμικά όργανα εν ευθέτω χρόνο πριν να παρουσιαστεί το σχέδιο προϋπολογισμού του 2016, λέμε. Δηλαδή, η συμφωνία που επετέθη μεταξύ των δύο κλάδων του προϋπολογισμού κατά την άποψή μας είναι κάτι αποδεκτό και θα πρέπει να υποστηριχθεί όπως έγινε και από τη Δευτέρα το βράδυ στην Επιτροπή Προπολογισμών με μεγάλη διαφορά. Λέγοντας αυτό κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αποσιωπήσω και κάποια μέτρια αποτελέσματα. 30 εκατομμύρια εδώ, 11 εκατομμύρια εκεί. Όσον αφορά αναδιπλώσεις ε, που θεώρησε ότι έπρεπε να, ε, να αφαιρέσει και από κάποιο κράτος μέλος με την απειλή περιστρόφου σχεδόν αυτές ε, οι μετριότητες ε, δεν ε, είναι προς τιμή τους. Και έχει και μανία το Συμβούλιο να καλύπτει τις ανάγκες των κρατών μελών. Και έλεγε ότι οφειλόταν το πλεόνασμα από την επαναξιολόγηση. Παρουσιάστηκε σχετικό κείμενο. Είμαι συνεισηγητής με τον κύριο Λεβαντόφσκι, στον οποίο θα αναθέσω να παρουσιάσει το κείμενο που θα ψήφιζα ε, αυθόρμητα ο Πρωθυπουργό, ο πρώην Πρωθυπουργό τελικά ήταν κάπω αντίθετο με όλα αυτά. Έχω πολλά πράγματα να πω, κυρία Πρόεδρε, αλλά θα τα αφήσω για τα δύο τελευταία λεπτά. Σα Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε εξαναγγείλει τον ε, συνεισηγητή σας. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Λεβαντόφσκι για τέσσερα λεπτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνουμε μια διαδικασία που ήταν δύσκολη για τον προϋπολογισμό 2014-2015. Ένα στοιχείο ήταν η διόρθωση του κανονισμού όσον αφορά τους ίδιους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κάτι που ζήτησε το Ευρωκοινοβούλιο. για πρώτη φορά δεν συμμετείχα στη συνδιαλλαγή αλλά πάντα υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις, προϋποθέσεις που τίθενται πέρσι αφορούσαν οι συνθήκες, της δημοσιονομικές προοπτικές ε, και τι θα γινόταν με τον προϋπολογισμό του 2014 φέτος. Μια άλλη ιδιαιτερότητα τονίστηκε οι πληρωμές βάσει των εθνικών συνεισφορών του ΦΠΑ και αυτό ε, περιέπλεξε τις διαπραγματεύσεις. Κάθε χρόνο υπάρχει ένα πρόβλημα. Ευρωπαϊκός προπολογισμό είναι σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν είναι εφεύρεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν είναι κάτι που γεννήθηκε από μόνο του. Είναι κάτι που υπέστη ε, αξιολογήσεις ε, αξιολογήσει από τα 28 κράτη-μέλη. Και γι' αυτό υπήρξε και απογοήτευση στις τελευταίες διαπραγματεύσεις. Αυτό το ποσό λοιπόν αμφισβητείται από τα κράτη-μέλη στην τελευταία φάση των διαπραγματεύσεων. Υπήρξε και μια άλλη συνθήκη ε, ιδιαίτερη, η θεμελιώδης αλλαγή της βάσης υπολογισμού του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος και του ΦΠΑ για κάποια κράτη-μέλη. Αυτό ήταν καλό σαν είδηση, για άλλες χώρες όμως ήταν κακά μαντάτα. Άλλοι πληρώνουν περισσότερα, άλλοι λιγότερα. Η Μεγάλη Βρετανία και η Φιλανδία ε, θα έχουν σημαντικό ποσό να καταβάλουν. Λοιπόν, αυτό το πρόβλημα οφειλόταν στα κράτη-μέλη και στο τέλος δεν μπόρεσαν να τοποθετηθούν τα κράτη-μέλη, αποφασίσουν ποια θα είναι η θέση τους. Περίμεναν από το Κοινοβούλιο όμως τη διαδικασία του κατεπήγοντος, την ε, επιταχυμένη διαδικασία. Σημειώσαμε αυτό το παράδοξο που υπήρχε. Από τη μία πλευρά ε, πατάνε στον, στο, στον γκάζι και από την άλλη στο φρένο. Συνεπώς, θεωρήθηκε και το θέμα των ιδίων πόρων σαν ένα στοιχείο της συμφωνίας. Τώρα έχουμε τον προπολογισμό για το 2014-2015 και θεωρούμε ε, θετικό επίσης ότι έγιναν και διορθώσεις του κανονισμού για τους ε, ίδιους πόρους. Υπάρχουν δύο διορθώσει για να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τα δημοσιονομικά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ανάγκη κοινοποίηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά καθυστερημένε πληρωμέ και είναι κάτι που απέρευσε από τον Ευρωπαϊκό προπολογισμό. Κάνουμε παρατηρήσει, δεν διαμαρτυρόμεθα. Κάνουμε κριτικέ παρατηρήσει. Όπω ήθιστε. αυτέ οι αλλαγέ των στατιστικών στοιχείων προήλθαν από τα κράτη-μέλη αυτά καθε αυτά μπορούν όμως καμιά φορά να διευκολύνουν τους ε, υπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λοιπόν, ε, υπάρχει μια ομάδα χωρών που τελικά ε, δεν δείχνει μεγάλη ευελιξία, δεν δείχνει καθόλου ευελιξία και αυτά τα κράτη-μέλη είναι τα πρώτα που ζητούν ταυτόχρονα περικοπές όσον αφορά τον προπολογισμό και ταυτόχρονα διεκδικούν και ανάπτυξη και αύξηση της απασχόλησης. Αυτό είναι κάτι που περιπλέκει πραγματικά την κατάσταση και γι' αυτό στη θέση του Κοινοβουλίου στην ομάδα υψηλού επίπεδου για τους πόρους λάβαμε υπόψη όλη την κατάσταση η πρόταση έγινε αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περασμένη εβδομάδα και ελπίζουμε ότι οι τυπικότητες, δηλαδή η ψηφοφορία στην Ολομέλεια θα γίνει αυτή την εβδομάδα. Ευχαριστώ κύριε και Ακούσαμε λοιπόν τους συζητητές και θα δώσω τώρα το λόγο στο Συμβούλιο του κύριο Μαντόβα. Έχετε 10 λεπτά. Αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και πιο λίγο χρόνο αν θέλετε. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, Αντιπρόεδρε Γεωργίευα, κυρίε και κύριοι, για μένα είναι μια τιμή να παίρνω το λόγο κατά τη διάρκεια τη Ολομελία για την συζήτηση που λαμβάνει η χώρα για την πολιτική συμφωνία που επετεύχθη στι 8 Δεκεμβρίου μεταξύ Συμβουλίου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2015 και το πακέτο των διεθνωτικών προπολογισμών για το 2014. Το Συμβούλιο ήδη επισημοποίησε την πρόθεσή του τις 12 Δεκεμβρίου και περιμένουμε, έχουμε κάθε πεποίθηση, ότι ποια θα είναι τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που προγραμματίστηκε για αύριο. Η συμφωνία επετέχθη σε ένα πλαίσιο διαπραγματευτικό, ιδιαίτερα περίπλοκο, λόγω των πολλών ερωτημάτων και θεμάτων που έπρεπε να αντιμετωπιστούν. Πιστεύω ότι ποτέ όπως φέτος δεν υπήρξαν τόσοι προπολογισμοί διορθωτικοί που έπρεπε να εγκριθούν Πιστεύω επίσης ότι ποτέ δεν έπρεπε να αντιμετωπίσουμε ένα τόσο υψηλό επίπεδο απλήρωτων λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτή είναι μια περίσταση που μας εμπόδισε και μας οδήγησε σε έντονο διάλογο και στο τέλος συμφωνήσαμε μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ακολουθήσουμε μια διαδρομή που τα επόμενα χρόνια θα μας επιτρέψει ε, την χρέωση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να την φέρουμε σε πιο αποδεκτά και βιώσιμα επίπεδα. Υπήρξαν διάφορες απόψεις για τη μείωση του επίπεδου των απλήρωτων λογαριασμών, των καθυστερημένων πληρωμών και στο τέλος πιστεύω ότι βρήκαμε έναν καλό συμβιβασμό. Είμαι συνεπώς σίγουρος ότι αν συμφωνήσει το Ευρωκοινοβούλιο ότι 3,5 δισεκατομμύρια παραπάνω δόθηκαν, πρικοδοτήθηκαν από το 2014 και ότι είναι θετικό και σημαντικό αποτέλεσμα για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα είναι καλό από τη στιγμή που τίθεται τέρμα στην ανάπτυξη του απαθέματος των απλήρωτων λογαριασμών και ταυτόχρονα δημιουργείται η βάση για μια σταδιακή απορρόφηση των απλήρωτων λογαριασμών τα επόμενα χρόνια. Όσον αφορά συγκεκριμένο το συνολικό ποσό για το 2015 αποτελείται αυτό από 2,818 δισεκατομμύρια ευρώ ε, που προέρχονται από το contingency περιθώριο 361 εκατομμύρια ευρώ που προέρχονται από τη χρήση των διαθέσιμων περιθωρίων όσον αφορά τα μέγιστα δαπανών του προπολογισμού του 2014 και τέλος άλλα 350 εκατομμύρια ευρώ που αφορούν τα ειδικά μέσα που προστίθενται στο contingency margin Οπότε στην επόμενη φάση θα πρέπει να βρεθεί μια συμφωνία μεταξύ θεσμικών οργάνων για να συμπεριληφθούν τουλάχιστον ε, στο μέγιστα των δαπανών. Πιστεύω ότι αυτό δείχνει ότι υπετεύχθη μια ισορροπία μεταξύ των δεσμεύσεων των δημοσιονομικών που δεσμεύουν τα κράτη-μέλη και των χρηματοδοτικών αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υλοποίηση των διαφόρων προγραμμάτων. Όσον αφορά τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2015, προβλέπονται 145,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε ε, αναλήψη υποχρεώσεων, συν 1, δηλαδή 1,8% παραπάνω σε σχέση με τον προπολογισμό του 2014, του προπολογισμού, 141,2 δισεκατομμύριο σε πιστώσεις πληρωμών, δηλαδή συν 1,6% παραπάνω σε σχέση με τον προπολογισμό του 2014, τροποποιημένου προπολογισμού. Λοιπόν, οι, αυτές, αυτά τα ποσά μας δίνουν επαρκή αποθέματα κάτω από τα μέγιστα του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 και έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορεί να έχει στη διάθεσή της επαρκή ποσά περιθώρια ελιγμών για να δράσει σε ενδεχόμενα πρόβλεπτα γεγονότα. Πιστεύω ότι το τρόπο ο προπολογισμό του 2015 θα εγγυηθεί τι αναγκαίε πιστώσει για εφαρμογή ευφυή e e και αποτελεσματική των νέων προγραμμάτων, λαμβάνοντα υπόψη ότι πρόκειται για τον δεύτερο ετήσιο προπολογισμό στα πλαίσια του νέου δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020. Ε, να δώσω κάποιο παράδειγμα, να επισημάνω ότι οι πληρωμές για το τίτλο 1α, ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και απασχόληση, όπου διατίθενται οι πόροι υπέρ της έρευνας, της κατάρτισης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που ε, έχουμε μια αύξηση 33% σε σχέση με τα 3,9 δις ευρώ σε συγκρίση με τον προβλησμό του 2014 ε, μαζί με τις αλλαγές που έγιναν και η πρικοδότηση για την πολιτική την εξωτερική Ευρωπαϊκής δέχτηκε μια αύξηση όσον αφορά τις πληρωμές περίπου κατά 8,5% αυξήσεις. Στις άλλες αυξήσεις επισημαίνουν τους πόρους που διατίθεται για τον τομέα του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων και των μεταναστευτικών ροών, καθώς και για την εποπτική υπηρεσία για τα δημοσιονομικά των ε, θεσμικών οργάνων. Όσον αφορά τη γεωργική πολιτική, ε, λάβαμε υπόψη τα αιτήματα των εμπόρων του τομέα και λάβαμε υπόψη και τις συνέπειες του εμπάργου του ρωσικού και θα δεχτούν συμπληρωματικές ε, υποστηρίξεις από ειδικά ποσά που θα Χωρίς να επηρεάσουμε όμως τα αποθέματα που θα είναι διαθέσιμα τα αποθέματα για ενδεχόμενα κατεπήγοντα που ίσως ε, συμβούν το 2015. Πιστεύω ότι αυτά τα αποτελέσματα θα πρέπει να αξιολογηθούν και υπό το φως του χρονοδιαγράμματος που ήταν εξαιρετικά ε, περιορισμένο και είχαμε στη διάθεσή μας για να καθορίσουμε τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσης για το επόμενο έτος έλειπε στη συνδιαλλαγή συμφωνία στις 17 Νοεμβρίου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια νέα πρόταση προπολογισμού για το 2015 και πρότεινε νέα συμβαστική πρόταση για ιδιωτικού προπολογισμού που εκκρεμούσαν για το 2014 στις 28 Νοεμβρίου. Παρ' όλα αυτά καταφέραμε να πετύχουμε μια συμφωνία στις 8 Δεκεμβρίου εν ευθέτω χρόνο για να μπορέσουμε να επιτρέψουμε και έγκριση αυτών πριν το τέλος του έτους και να αποφύγουμε την προσφυγή στα δεκατημόρια τα, προσωρινά για το 2015. Οι διαπραγματεύσεις λοιπόν ήταν εντατικότατες, πετύχαμε μια συμφωνία και αυτό είναι πολύ θετικό μήνυμα που στέλνουμε όσον αφορά τη δυνατότητα που έχουν τα δύο θεσμικά μας όργανα να συνεννοούνται ε, και να μπορούν να συγκεράσουν τα συμφέροντα των πολιτών μας. Ε, θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τα επιτευχθέντα αποτελέσματα και ευχαριστώ όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στις διαπραγματεύσεις. Κυρίως θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Αρτουή και τους εισηγητές κύριε Γκαρτζιαμπραλ, Χολμάιερ και Ντεπρέ οι οποίοι προσπάθησαν, έκαναν προσπάθειες διαπραγματεύσεις, είχαν επικοδομητική στάση και πνεύμα συνεργασίας όταν απαιτείται. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, Αντιπρόεδρε, κυρία Γεωργίευα και την ομάδα σας ε, διότι με τη σειρά σας διευκολύνατε με μεγάλη αμεροληψία τη θετική ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Κλείνω εκφράζοντας την πεποίθησή μου ότι η συμφωνία που πετέφθη με το Κοινοβούλιο αντιπροσωπεύει μία απάντηση πλήρως συνεκτική που ταιριάζει με τις τρεις κρίσιμε προκλήσει που περιμένουν του χρόνου. Να συνεχίσουμε να μειώνουμε ε, τους του λογαριασμού, να μην υπονομεύουμε την προσπάθεια που καταβάλουν τα κράτη-μέλη για την εξυγίανση των δημοσιονομικών του εθνικό επίπεδο, να δώσουμε τα απαραίτητα ποσά και κίνητρα για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης ε, που είναι επωφελής για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε. Θα λάβει τον λόγο η Επιτροπή. Η Επίτροπος Γεωργίευα. Δέκα λεπτά έχετε στη διάθεσή σας. Φυσικά μπορείτε να είσαστε πιο σύντομοι. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε για την ευκαιρία που μου προσφέρετε να προσφωνήσω τους Ευρωβουλευτές πριν από την ψηφοφορία αύριο στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού για το 2014, τον προϋπολογισμό του 2015, σχέδιο προϋπολογισμού 2015 και την τροποποίηση για τον κανονισμό 1150. Όλοι νομίζω συμφωνούμε επ' αυτόν ότι ήταν πολύ δύσκολες οι διαπραγματεύσεις για αυτά τα θέματα. Είναι το πρώτο έτος του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου που τίθεται σε εφαρμογή αυτά τα οποία σχεδιάστηκαν για πρώτη φορά στο τέλος τέλος. Και είναι και η χρονική συγκυρία που έπρεπε να εξευρεθούν τρόποι και μέσα και λύσεις να σταθεροποιηθεί το επίπεδο των μη εκτελεστησών πληρωμών και όπου πολλά από τα κράτη-μέλη μας αντιμετωπίζουν μια πολύ δύσκολη ε, δημοσιονομική κατάσταση όμως εργαστήκαμε πάρα πολύ σκληρά να βρούμε την σωστή οδό προς ένα συμβιβασμό και μια συμφωνία. Θέλω να ευχαριστήσω το δημοσιονομικό σκέλος της αρμόδιας επί του προϋπολογισμού δημοσιονομικών δηλαδή αρχής για ένα <clears throat> σταθερό αξιόπιστο προϋπολογισμό που διασφαλίζει τη συνέχεια και την προβλεψιμότητα. Αλλά πιο σημαντικό απ' όλα στέλνει ένα μήνυμα στους πολίτες ότι παρόλες τις διαφορές και τις δυσκολίες μπορούμε να καταλήξουμε και να βρούμε μια λύση, κοινή λύση όλοι μας, ε, στοχεύοντας προς ένα κοινό στόχο. Και ευχαριστώ πολύ εσάς ε, Πρόεδρε για τον ηγετικό ρόλο, την πρωτοβουλία που είχατε αναλάβει στις διαπραγματεύσεις. Φυσικά ευχαριστώ και τους εισηγητές, την κυρία Καρδιασάβαρ, την κυρία Χολμάιερ και α, που είναι εκεί σωστά και τον κύριο Ντεπρέ, ε, Ντεπρέ επιτέλους επίσης και φυσικά τον πρώην συνάδελφό μου επίτροπο, πρώην επίτροπο Λεβαντόφσκι, τώρα ευρωβουλευτή, για όλα όσα έπραξε κατά την προηγούμενη ιδιότητα του που μας βοήθησε να καταλήξουμε σε αυτή τη συμφωνία τελικά και θέλω να ευχαριστήσω φυσικά και την Ιταλική Προεδρία, τον ε, Υπουργό Παντουάν, που προσήλθε σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή και εργαστήκατε άοκνα όλοι σας για να συνοδεύσετε και να παρακολουθήσετε αυτή τη διεργασία. Και έχουμε τώρα μια λύση που ελπίζω ότι θα υπερψηφιστεί αύριο, διότι είναι μια θετική έκβαση των διαπραγματεύσεων. Φυσικά εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύουμε ότι αυτό που αρχικά είχε προταθεί ήταν αξιόπιστο και Αλλά μπορούμε να δεχθούμε και αυτό που τροποποιήθηκε τώρα από την αρχική μας πρόταση και όπως πολλοί από εσά είπατε είναι κέρια σημασία να εξυπηρετήσουμε τα προγράμματά μας, να λειτουργήσουν τα προγράμματα υπέρ των πολιτών μας. Πρώτα απ' όλα να πω δύο λόγια αν επιτρέπετε για το 2014, το, τα σχέδια διορθωτικών προπολογισμών δηλαδή σχετικά με το 2014. Ένα ιδιαίτερα σκληρό έτος υπό το δημοσιονομικό πρίσμα, διότι ταυτόχρονα αντιμετωπίσαμε πίεση για των πληρωμών της προηγούμενης προγραμματικής περίοδου που έφτασαν στο τελευταίο του έτος και την ανάγκη να υπάρξει ένα νέο πλαίσιο για τα πολιετή δημοσιονομικά πλαίσια και την ανάγκη για τις πρόσθετες, ε, ε, ε, τη, διασφάλιση των πρόσθετων κονδυλίων για το 2014, ιδιαίτερα με τον διορθωτικό προϋπολογισμό 3, την κινητοποίηση δηλαδή των περιθωρίων και την μέγιστη, βέλτιστη χρήση των δυνατοτήτων που υπήρχαν κέρια σημασίας για την ε, ε, ευδοκίμηση των διαδικασιών και θα έλεγα επίσης προλυαίνοντας το έδαφος και για τον προπολογισμό 2015 ακούσαμε την αξιολόγηση των αριθμητικών μεγεθών. Να προσθέσω τρεις σύντομες παρατηρήσεις επ' αυτών. Πρώτον, εποφελούμεθα επιπλέον από κάποιες ε, νέες χρήσεις ε, και όσον αφορά ε, κονδύλια που μετατίθενται από το 2014 προς το 2015. Βέλτιστη χρήση όσον αφορά τα συνολικά κονδύλια για τα χρήματα για την πληρωμή λογαριασμών που θα φτάσουν στα 4,4 δις ε, το 2015. Από αυτά θα έχουμε 400 ε, εκατομμύρια πρώτο, στο, πρώτο, ε, στο πρώτο κεφάλαιο. Θα έχουμε 7 δισεκατομμύρια, 60 εκατομμύρια επιπλέον για την ενίσχυση διεθνών προγραμμάτων, για την δυνατότητα να συνδράμουμε όλους όσους έχουν ανάγκη για τον προϋπολογισμό του 2015. Επιτρέψτε μου να σκιαγραφίσω αυτά που θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα αξιόλογα σε σχέση με αυτή τη συμφωνία. Πρώτον, επικεντρώνεται στις επενδύσεις σας, στις πολιτικές προτεραιότητες που έχουμε εμείς θεσπίσει τονίζει αυτό που πρέπει να γίνει για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και ιδιαίτερα τα 350 δισεκατομμύρια, 315 δισεκατομμύρια που παρουσιάσαμε ως πρόγραμμα επενδύσεων ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζεται η σημασία τους. Επίσης σε σχέση με τον προπολογισμό 2014 έχουμε επαρκή αλλά, μετριοπαθή αλλά επαρκή αύξηση που θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τις πιέσεις που προανέφερα για την αύξηση σε σχέση με τις ε, υποχρεώσεις πληρωμών για 2,6 δις για τις πληρωμές 1,6% δηλαδή 2,2 δις που θα διατεθούν. Επιτρέπει επιπλέον να διαθέσουμε στην κατηγορία Α περισσότερα χρήματα και επίσης και στην κατηγορία 4 όπου οι πιέσεις είναι ιδιαίτερα ισχυρές και όπως ανέφερε η Προεδρία καταφέραμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των γεωργών που επλήγησαν από την απαγόρευση εξαγωγών των προϊόντων του στη Ρωσία καθώς επίσης και για τα κατακτοκομικά χωρίς ε, να υπάρξει ανάγκη να χρησιμοποιηθεί το αποθεματικό κρίσεων. Επίσης έχουμε, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο και πρέπει να το αναγνωρίσουμε, μια πολύ υγιή ανάπτυξη όσον αφορά την αναλογία μεταξύ υποχρεώσεων και πληρωμών για το 2014 και 2015. Σαν αποτέλεσμα αυτών που κάναμε είναι 97% αυτή η αναλογία σε σχέση με ε, το 89% που ίσχυε για αυτή την αναλογία κατά το παρελθόν. Τι σημαίνουν όλα αυτά. Σημαίνουν ότι θα είναι πιο εύκολο να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες και τα προβλήματα ε, όσον αφορά την υπερβολικά μεγάλη ταχύτητα πολλές φορές των εξελίξεων και των διαδικασιών. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από το αίτημα του Κοινοβουλίου που έγινε δεκτό από το Συμβούλιο να υπάρξει ένα, ένας προγραμματισμός πληρωμών, διότι αυτό θα οδηγήσει σε αηφορία, σε βιωσιμότητα και ήδη η Λετωνική Προεδρία, η επόμενη δηλαδή Προεδρία, συζητεί και ε, με ιδιαίτερα σοβαρό τρόπο αντιμετωπίζει το θέμα αυτό. Συναντήθηκα με τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Εξωτερικών που θα είναι αρμόδιος υπουργός για την ε, Λετωνική Προεδρία κατά την, το επόμενο εξάμεινο. Το πρόγραμμα ε, πληρωμών είναι για μας ένα εργαλείο, ένα μέσο για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτά τα οποία βιώσαμε εφέτος και αντιμετωπίσαμε ως ζήτημα σε σχέση με τις μη εκτελεστήσεις πληρωμής, πλη, μη εκτελεστήσεις πληρωμών. Σε αυτές τις διαπραγματεύσεις ε, συμφωνήσαμε να διαφωνούμε και αφήσαμε το θέμα ανοιχτό. Ιδιαίτερα όσον αφορά τις οροφές για το 2014 που θα πρέπει να εξεταστούν λέγοντας όμως ότι δεν είναι η τελική συμφωνία αυτή. Έπρεπε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση ελπίζοντας ότι θα, μπορούσε, θα μπορέσει να ολοκληρωθεί. Τώρα, στην αντιμετώπιση του θέματος των ε, μεγάλων προσαρμογών που έπρεπε να γίνουν όσον αφορά το GNI 9,5 δις σε προσαρμογές που κάποια κράτη-μέλη τα εξέπληξαν και τα ευνηδίασαν έχουμε μια περιορισμένη πρόταση περιορισμένου εύρους για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Οκτώ κράτη-μέλη έχουν, ε, ε, όπως προβλέπει η τροπολογία αυτή, ε, να τοποθετηθούν. Αναμένω ότι θα γνωμοδοτήσει το Κοινοβούλιο επ' αυτού, ελπίζοντας θα γνωμοδοτήσει θετικά. Ολοκληρώνω με τρεις παρατηρήσεις. Πρώτον, έχουμε ένα προϋπολογισμό τώρα. Πρέπει να κάνουμε τη βέλτιστη χρήση αυτού του προϋπολογισμού που έχουμε στα χέρια μας. Αυτό είναι η ανώτατη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να επικεντρωθεί στα αποτελέσματα, βέλτιστα αποτελέσματα όσον αφορά την ποιότητα των ε, πληρωμών. Και για τη συνάντηση και τη δράση των ε, υψηλών αξιωματούχων ε, για τους ιδίους πόρους ε, με πολύ πραγματικά κέριο έργο, ε, κέρια σημασίας για την ολοκλήρωση των στόχων επιτελείται. Και τέλος αλεξίσου σημαντικό, βρισκόμαστε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ακούσατε σε σχέση με το νέο πρόγραμμα εργασίας, έχουμε στεναρή δέσμευση για να υπάρξει ευθυγράμμιση των προτεραιοτήτων μας όσον αφορά τον προϋπολογισμό ώστε να καταδείξουμε στους πολίτες μας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει σωστά τη δουλειά της εκεί όπου έχει σημασία κάνει τη δουλειά της σωστά προς όφελος των πολιτών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Επιτρόπε και επόμενος ομιλητής από πλευρά τη Επιτροπή Περιφερειακής ανάπτυξη για δύο λεπτά έχει το λόγο ο κ. Ολμπρίχτ. Όχ, από Σας ευχαριστώ. Σήμερα λοιπόν ε, συζητάμε τον προπολογισμό πριν από την ψηφοφορία. Στην πραγματικότητα όμως εκφράζουμε μεγάλη ε, ικανοποίηση για το γεγονός ότι έχουμε πετύχει συμβιβασμό. Θα πρέπει να είμαστε λοιπόν ικανοποιημένοι και θα πρέπει η ικανοποίηση αυτή να ενδοθεί ως κατησχετικό. Φυσικά είναι καλύτερο να υπάρχει ε, προπολογισμό παρά να υπάρχουν τα 12 αρτημόρια. Είναι σαφέ. Είναι πολύ πιο σωστό να υπάρχει προπολογισμό. Ξέρουμε επίση ε, τι θα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει, αλλά θα πρέπει να έχουμε συνείδηση του ότι οι διαπραγματεύσει ήταν πάρα πολύ δύσκολε, εξαιρετικά δύσκολε και το τόνισε η κυρία Επίτροπο άλλωστε αυτό. Κάποια στοιχεία τώρα πολύ χαρακτηριστικά αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων αυτών. Καταρχάς, ότι δεν μπορέσαμε να επικεντρωθούμε στον προπολογισμό του 2015, αλλά προσπαθήσαμε μάλλον να κλείσουμε τα χάσματα του 2014. Μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσαμε να καλύψουμε τα κενά. Συζητήσαμε το θέμα, δηλαδή να δούμε πώς μπορούμε να αποφύγουμε μια καταστροφή το 2014 ε, έγινε μια σοβαρή συζήτηση όσον αφορά τις συνέπειες που θα, συνέ... θα σήμαινε αυτό για τον προπολογισμό του 2015. Ήταν άνευ προηγουμένου αυτή η κατάσταση, διότι τα προηγούμενα έτη η συζήτηση όσον αφορά το έτος 2015 ήταν λεπτομερέστατη, είχε ξεκινήσει καλά εκ των προτέρων πολύ πριν και το έτος 2014 και το έτος 2015 για την περιφερειακή πολιτική είναι πολύ σημαντικά έτη. Η κυρία Επίτροπος υπογράμμισε ότι αυτά τα δύο χρόνια σύμφωνα με, με τον κανόνα νήσιν 2 ε, είναι χρονιές ε, για το κλείσιμο των λογαριασμών. Δηλαδή, με άλλα λόγια, όλες, ε, όλα τα αιτήματα για πληρωμές θα καταφτάσουν το 2014 και το 2015. Και όλοι γνωρίζουμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα. Για να το πούμε αλλιώς, η ε, ικανοποίησή μα όσον αφορά τι διαπραγματεύσει και τον προπολογισμό είναι σχετική ικανοποίηση. Πρέπει το ερώτημα κατά πόσο το σύστημα είναι βιώσιμο. Σα ευχαριστώ κυρία Όλμπριχτ και τώρα εξ ονόματο ε, των ομάδων ο πρώτο ομιλητή για δύο λεπτά είναι ο κύριο Φερνάντο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Επίτροπε, κύριε εκπρόσωπε του Συμβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ όλους όσους παρενέβησαν, διότι θεωρώ ότι η Ένωση, η ο ενωμένο τρόπος με τον οποίο εργαστήκαμε και το σθένος επέτυχε αυτό τον, αυτή τη συμφωνία για τον προϋπολογισμό και διορθωτικούς προϋπολογισμούς του 2014 και για τον προϋπολογισμό του 2015. Είναι θεμελιώδου σημασία και το πρόγραμμα πληρωμών για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέμε πληρωμές ενώ είναι οφειλές, γιατί για οφειλές πρόκειται. Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως η συγκεκριμενοποίηση των προτεραιοτήτων μας για την απασχόληση και τις απασχόλησης, αυτή η συμφωνία δίνει τη δυνατότητα να σταθεροποιηθεί το χρέος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μπορέσει να λειτουργήσει ο προπολογισμό. Έτσι το 2014 τέσσερα δις επιπλέον ε, που χρειαζόντουσαν και διασφαλίστηκαν για να καλυφθεί το επίπεδο των μη εκτελεστησών πληρωμών με έκτακτες δυνατότητες εσόδων ε, το 2014 που απέρεαν από πρόστιμα. Χωρίς αυτή τη συμφωνία τα κράτη-μέλη θα έπαιρναν ε, αυτά τα χρήματα όσον αφορά από τους εθνικούς προϋπολογισμούς, πράγμα το οποίο θα ήταν απαράδεκτο, επειδή ήταν όχι μόνο υψηλό το επίπεδο αυτών των ποσών όπως αναφέρθηκε, αλλά και η πίεση των κρατών μελών. Επίσης, καταφέραμε οι περικοπές του Συμβουλίου που είχαν προταθεί να ελαχιστοποιηθούν οι περικοπές αυτές. Επίσης ενισχύσαμε τις δεσμεύσεις όσον αφορά τα προγράμματα για την απασχόληση και την δημιουργία ε, επενδύσεων. Η ε, ευρωπαϊκή αλληλεγγύη ενισχύεται επίσης ε, όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια που χορηγείται. Το 2015 όπως συμφωνήθηκε σε σχέση με την Επιτροπή και το Συμβούλιο πρέπει να υπάρξει ένα πρόγραμμα για να αντιμετωπίσουμε τους λογαριασμού και που, που δεν έχουν έχουν εκτελεστεί. Η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση πρέπει να είναι εξίσου αυστηρή με τον εαυτό της όπως είναι αυστηρή με τα κράτη-μέλη και να, δεσ... να υλοποιεί τις δεσμεύσεις της όσον αφορά το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ, λέει πρόεδρος. Επόμενος ομιλητής για δύο λεπτά είναι ο κύριος Γκάιερ. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Κύριε Φιμπουργέ Ντέλοβα, κύριε Αντιπρόεδρε ε, Γκίεβα, θα μπορώ να πω και εγώ εξ ονόματος των Σοσιαλδημοκρατών ότι και εγώ συγχαίρω ιδιαίτερα στην Προεδρία του Συμβουλίου γιατί δεν μπορούμε να το τονίσουμε αρκετά ότι αν ε, σε μια τέτοια φάση κρίσιμη το Συμβούλιο χρειαζόταν 21 μέρες για να βρει την κοινή θέση καν η οποία στη συνέχεια μετά τις πρώτες διαπραγματεύσει, επειδή δεν μπόρεσε να περάσει αυτή η κοινή θέση, έπρεπε να ξαναξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις. Ο μόνος που θα πρέπει να συγχαρούμε είναι την Ιταλική Προεδρία, που κατάφερε να κρατήσει την, ε, το Συμβούλιο. Αυτό που ζούμε με το Συμβούλιο είναι φάση ψυχοθεραπείας. Η πρώτη φάση ε, θεραπείας είναι η άρνηση. Την περάσαμε αυτή την άρνηση που, τη φάση που το Συμβούλιο αρνούταν τους ε, αριθμούς, τα ποσά τα οποία ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είχαμε και τη φάση της αντίστασης και αυτό το περάσαμε. Το Συμβούλιο λέει πλέον ότι ναι, είμαστε διτεθειμένοι να δώσουμε στην ε, Ευρωπαϊκό Προπολογισμό νέο χρήμα, γιατί δεν μπορούμε να αρνηθούμε το χάσμα των πληρωμών. Πολύ καλό και αυτό. Και τώρα είμαστε στη φάση της θεραπείας. Πρέπει να έρθει και η θεραπεία. Και χάρηκα που άκουσα από εσάς, κυρία Αντιπρόεδρε, ότι είστε ήδη σε διάλογο με τη Λετωνική Προεδρία. Γιατί η Λετωνική Κυβέρνηση θα πρέπει να είναι εκείνη η οποία θα τα εφαρμόσει όλα αυτά για το σχέδιο πληρωμών. Θα πρέπει να δώσει ζωή στο σχέδιο πληρωμών. Εμεί από την πλευρά τη Επιτροπή Προπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν μπορούμε να φανταστούμε τίποτε άλλο παρά τακτική αναφορά από εσάς κύριε Αντιπρόεδρε για το πώς ε, θα συνεχιστούν οι πληρωμές. Ελπίζω να επαληθευτούν οι προβλέψεις και ότι θα φτάσουν τα χρήματα προκειμένου να απαλληλθεί αυτή η κρίση πληρωμών. Δεν είμαι και πολύ αισιόδοξο να σας πω την αλήθεια. Θα πρέπει να φροντίσουμε προκειμένου στο μέλλον ε, το Συμβούλιο στις διαπραγματεύσεις του να κάνει τα λόγια του πράξης. Είδαμε λοιπόν ότι μπορούμε να είμαστε πάρα πολύ υπομονετικοί και δεν πρόκειται να αρκεστούμε στα λόγια στο μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για δυόμιση λεπτά ο κύριος Κιόλμελ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαιρετίζω την Επίτροπο κυρία Γεωργίευα, τους εκπροσώπους του Συμβουλίου και φυσικά ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχαν στην εκπόνηση αυτών των εγγράφων και προτάσεων παρότι εμείς από την ε, ομάδα μας ε, με το αποτέλεσμα δεν είμαστε καθόλου ικανοποιημένοι. Αυτή την εβδομάδα θα συζητήσουμε μια ολόκληρη δέσμη μέτρων που πρόκειται να εγκριθούν και πρόκειται για διαφορετικούς συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς για το 2014 Αφενός πρόκειται για την ε, βοήθεια σε περιπτώσεις καταστροφών, θεομηνιών, αλλά και προσαρμογές. Και εγκρίνουμε αυτά χωρίς επιφύλαξη. Όμως πρόκειται επίσης και για την χρηματοδότηση εκκρεμουσών πληρωμών. Αυτό είναι σημαντικό και έχει υπαρξιακή σπουδαιότητα. Όμως αυτές, αυτοί οι συμβιβασμοί που εκπονήθηκαν δεν επαρκούν. Πόρο απέχουν από το να επαρκούν. Τέσσερα δις προβλέπονται επιπλέον για αυτό το έργο. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρέη 23 δις και μάλιστα υπό τη μορφή μη ε, λογαριασμών και πληρωμών που εκκρεμούν. Χρέη που πρέπει να πληρωθούν. Εμείς ως CCR ως ομάδα άρα απορρίπτουμε αυτούς τους, ε, αυτά τα αιτήματα. Αν δούμε τον προϋπολογισμό του 2015 πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι στην έναρξη του έτους θα έχουμε 20 δις χρέη ήδη και μέσω αυτού τα διαθέσιμα ποσά για πληρωτές από 141 δις θα μειωθούν σε 121 δις αυτόματα. Ταυτόχρονα όμως έχουμε προβλέψει όσον αφορά 144 δις υποσχέσεων πληρωμών, δεσμεύσεων για πληρωμές, διαρωτώ με εγώ και ερωτώ όλους σας πώς, μπορεί αυτοί, πώς μπορούν αυτοί οι λογαριασμοί να είναι σωστοί. Τολμώ να σας πω ότι δεν είναι σωστοί και δεν μπορούν να λειτουργήσουν όλα αυτά εκτός αν υπάρξουν νέες ρυθμίσεις και νέοι κανόνες που θα εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα έλεγα ας μην προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι τέλο. Και μια και δεσμεύτηκαν πληρωμές που δεν είμαστε ικανοί να εκτελέσουμε πάνω από από 200 δις, τότε η κατάσταση καθίσταται ακόμα πιο δραματική. Η δημοσιονομική διαδικασία είναι πολύ περίπλοκη. Κάνουμε λόγο για ειδικά αποθεματικά, γενικά αποθεματικά, μέσω ελαστικότητας, on top ή μη on top, όλα αυτά δεν είναι καθόλου διάφανα και μου υπενθυμίζουν περισσότερο αυτό το οποίο είπε ο George Orwell που είχε πει στο Newspeak κατά το παρελθόν ότι η πολιτική ομιλεί με τέτοιο τρόπο ώστε οι πολίτες να μην καταλαβαίνουν γρή. Και κάτι τελευταίο βλέπω σε σχέση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 141 δις το κοινοβούλιο λέει 140, το κοινοβούλιο 146 ε, καταλήξαμε τώρα, δια... Ε, καταλήγει πρόεδρος και λέει έληξε ο χρόνος σας, σας ευχαριστούμε, έληξε ο χρόνος σας κύριε σας ευχαριστούμε και ζητώ συγγνώμη που σας διέκοψε αλλά θέλω να ολοκληρωθεί η συζήτηση έγκαιρα. Επόμενος αγορητής, η πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμών, ο πρόεδρος Μισελ Ακτουή της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, να ευχαριστήσω την συγκήτρια την κυρία Γκαρδιαζαμπάλ, καταρχάς τον κύριο Αλμαΐρ, τον κύριο Ντεπρέ, να ευχαριστήσω την κυρία κυρία Γεωργίευα, να ευχαριστήσω την Ιταλική Προεδρία και συγκεκριμένα τον κύριο Σανίδο, τον πρέσβη. Είμαστε στις παραμονέ της ψηφοφορία του προπολογισμού μας. Θα ήθελα να εκφράσω ε, με ένα παράπονο και μια ελπίδα. Για τη διαδικασία δημοσιονομική έχω παράπονο. Τις τρεις εβδομάδες της συνδιαλλαγής, εκτός από τον, Γάλλο, από τον Ιταλό Υφυπουργό, δεν μπορούσαμε να ανταλλάξουμε με τους συνομιλητές μας ε, των κυβερνήσεων ε, κουβέντα. 28 ε, δεν έστειλαν ε, υπουργό. Περιμέναμε την 21η μέρα, τελευταία μέρα τη συνδιαλλαγή, ούτω ώστε το Συμβούλιο επιτέλου να μορφωστοποιήσει τι προτάσει του. Δυστυχώ ήταν απαράδεκτε. Η σώρευση των οποίων των λογαριασμών στο γραφείο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή των λογαριασμων στο γραφειο τη ευρωπαικη επιτροπη πλησιαζει στα 30 δισεκατομμύρια είναι σοβαρή απόκληση που δυσκολεύει πάρα πολλού εμπορευόμενου και υπονομεύει ε, την. Ε, αξιοπιστία Ευρωπαϊκής Ένωσης και ήταν παράδοξη στάση του Συμβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2014 είχε απρόβλεπτους πόρους 5 δισεκατομμύρια που προέβηναν από, από ε, πρόστιμα και τόκους, υπερημερίε και θέλαμε προτεραιότητα να πληρωθούν οι πιο επίγοντε λογαριασμοί. Το ζητήσαμε και αρνήθηκε το Συμβούλιο, το ζήτησε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εξεπλάγει από τον αυτισμό των κυβερνήσεων, των εθνικών κυβερνήσεων, που αρνούνται να υπομισθούν τι ευθύνε του και να ανταποκριθούν στι υποχρεώσει, ενώ δεχτήκαν τι αναλήψει υποχρεώσεων. Έλλειψη Υπήρχε έλλειψη των Υπουργών από τι διαπραγματεύσει. Αρνήθηκαν να πληρώσουν τα χρεωστούμενα. Να επενθυμίσουμε ότι οι πληρωμέ είναι η συνέπεια, η μηχανική συνέπεια των προηγούμενων αποφάσεών του. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που ζητούσαμε δεν θα μπορούσε παρά να ζητάμε τη σταθεροποίηση του χρέου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιμένουμε για το 2014 4 δισεκατομμύρια, 700 εκατομμύρια και πήραμε τελικά 3,5 δι. Για το 2015 περιμέναμε 2,3 δι και τελικά μα δόθηκαν 1,3 δι. Συνολικά 4 δι 800 εκατομμύρια αντί 7 δι. Άρα είναι σαφές αγαπητοί συνάδελφοι ότι τα ποσά επί των οποίων σφαγίσαμε τη συμφωνία μας, δεν ρυθμίζουν τα πρόβλημα. Αλλά αυτό που δημιουργεί την εμπίδα μου είναι ότι διάφοροι δεσμεύτηκαν να εφαρμόσουν μια δικασία εξυγίανση ε, του μεγάλου αυτού χρέου που δημιουργείται από του απλού λογαριασμού. Πρέπει να γνωρίζουμε επακριβώ αυτά τα ποσά στη 31 Δεκεμβρίου του 2014 και θα πρέπει να συμφωνήσουμε τι μπορεί να θεωρηθεί σαν λογικό και βιώσιμο ποσό. Ε, η εξυγίανση θα αφορά τη διαφορά μεταξύ των δύο και θα πρέπει να ρυθμιστεί το ταχύτερο δυνατόν. Αν το προβλεπόμενο ραντεβού το 2016 για την αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου ε, θα πρέπει ίσως να μας κινητοποιήσει από την αρχή του έτους 2015 για να κάνουμε τα δέοντα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you. Our next speaker for... Ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό η κυρία Νίη Ριάδα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και τους συζητητές, αλλά και τον Πρόεδρο για όλο τους ε, το έργο. Είναι πάρα πολύ σαφές ότι ο προπολογισμός του 2015 μας δείχνει ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, ένα τεράστιο χάσμα ανάμεσα στην Ευρώπη των πλουσίων και την Ευρώπη των φτωχών δεν πρόκειται να καλυφθεί αυτό το χάσμα γιατί ακολουθούμε πολιτικές λιτότητες. Επανειλημμένα έχω τονίσει την νικτρή κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο λιευτικός τομέας στην Ιρλανδία και με τις περικοπές έχει χειροτερέψει ακόμα η κατάσταση. 900 εκατομμύρια ευρώ θα τους βγάλουν από την κατηγορία 2. Πώς μπορεί ο κόσμος ο ευάλωτο στην κοινωνία μα να επιβιώσει. Πρέπει να βοηθήσουμε εκείνου που δεν μπορούν οι ίδιοι να αυτοβοηθηθούν. Επίση, η ανθρωπιστική βοήθεια μειώθηκε σε σχέση με το 2014 ακριβώ ε, λόγω των περικοπών στον τίτλο 4. Έχω αγανακτήσει. Ε, για τις ε, τόσο μεγάλες διαδραστικές περικοπές. Ε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια και την επίγουσα βοήθεια, ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε τη ε, δυνατότητα να αντιμετωπίζουμε τις θεομηνίες και την εκτρή κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι πρόσφυγες. Όταν έρθει ο προπολογισμό τον Ιανουάριο, το σχέδιο διορθωτικού θα πρέπει οπωσδήποτε να επηρεάσει τις κατηγορίες 1α και 1β να αποκατασταθούν τα ποστά το συντομότερο. Ευχαριστώ κυρία Νιρέντα. Α, νομίζω ότι ε, έχει μια μπλε κάρτα κάποιος συνάδελφος. Ε, δέχεστε την ερώτηση. Για 30 δεύτερα παρακαλώ, η κυρία Μόρη. Θα ήθελα να μάθω από την συνάδελφο, μιας και ζήτησε να αυξηθούν οι επιδοτήσεις και για τους μετανάστες στα κέντρα υποδοχής αν έχει δει τι συμβαίνει στην Ιταλία και τι απάτες ε, γίνονται, τώρα ήρθε στην επιφάνεια ένα νέο σκάνδαλο ότι και τα κόμματα της δεξιάς και τα κόμματα της αριστεράς έκλεψαν τα χρήματα που προοριζόντουσαν για τους φτωχούς και προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν την τραγική κατάσταση. Λοιπόν, πριν ζητήσετε λεφτά, δεν κοιτάτε να δείτε πού πήγαν τα προηγούμενα. Ευχαριστώ και 30 δεύτερα για την απάντηση. Παρακαλώ. Ναι. Δεν ε, γνωρίζω όλες τις λεπτομέρειες. Θα πρέπει πρώτα να διευκρινιστεί η κατάσταση, να δούμε τι συνέβη. και να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και για το από πού προέρχονται τα χρήματα αλλά και σε ποιον απευθύνονται. Ελπίζω να Κατάλαβατε αυτό που σας είπα. Ναι, ευχαριστώ. Δεν έχετε το λόγο. Είχατε 30 δεύτερα για να κάνετε την ερώτησή σας και απάντησε η ομιλήτρια. Για τρία λεπτά τώρα ο κύριος Τάραντ, παρακαλώ. Thank you, Madam President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην πολιτική μας ομάδα αναγνωρίζουμε την εξαιρετική δουλειά που έκανε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμών και οι συγγητές Δεχόμαστε και την ε, κατάληξη στην οποία οδηγηθήκαμε, η οποία δυστυχώς ε, ε, δεν είναι καλή, αλλά είναι ίσως καλύτερη από άλλες χρονιές. Νομίζω όμως ότι η συμφωνία αυτή δεν επιτρέπει τη σταθεροποίηση στον τομέα των πληρωμών. Όπως είπε ήδη και ο κύριος Ντεπρέ, είχαμε τρεις στόχους, τρεις στρατηγικούς στόχους Πρώτον, σταθεροποίηση στην κατάσταση των πληρωμών. Αποτύχαμε. Οι απλήρωτοι λογαριασμοί σωρεύονται. Δεύτερον, διαφοροποίηση για τα ειδικά μέσα. Και εκεί αποτύχαμε γιατί απόφαση δεν υπάρχει. Τρίτον, έπρεπε να έχουμε εμείς ε, ένα πρόγραμμα για να μπορέσουμε να μειώσουμε γενικά τις έκτακτες χρηματοδοτήσεις και αυτό ακόμα ε, δεν το πετύχαμε. Η κυρία Γουαρντασάμπαλ είπε ότι δεν συμφωνεί με τους αριθμούς αλλά θα στηρίξει την πρόταση. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί πρέπει να στηρίξουμε αυτή τη συμφωνία και γιατί να φοβόμαστε τόσο πολύ τα προσωρινά 12 Αντίθετα, θα πρέπει να στηρίξουμε τη μέθοδο των προσωρινών 12 τιμωρίων, διότι μόνο αυτή η μέθοδος θα πιέσει τις κυβερνήσεις και το Συμβούλιο να κατανοήσουν το βάθος του προβλήματος και ίσως να κάνουν και κάτι για να το λύσουν. Έχω γενικά πάρα πολλά να πω δεν θα τα πω όμω, γιατί όσοι ασχολούνται με τον προϋπολογισμό τα γνωρίζουν. Αλλά ε, ε το τέλος της ε, τρίτης, τρίλεπτης ομιλίας μου θα είμαι λίγο συναισθηματικό. Αν απορρίψουμε τον προϋπολογισμό. Σκεφτείτε το αυτό. Θα έχουμε για κανένα δυο μήνε προσωρινά δωδεκατημόρια και θα έχουμε μια νέα κατάσταση για τη σύνθεση του προπολογισμού αμέσω μετά. Αυτός δεν είναι και ο πραγματικός ρόλος του Κοινοβουλίου σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Γιατί όπως είπε και ο Λέων Αρκοέν δυστυχώς οι καλοί χάσανε, δυστυχώς η συμφωνία είναι χάλια. Ευχαριστώ κύριε Τάραντ, μισή λεπτό, τσάνι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω ότι η συμφωνία η οποία έγινε την τελευταία στιγμή ήταν η μοναδική ευκαιρία να έχουμε πραγματικά ένα, προ, ένα προϋπολογισμό βιώσιμο εκτός 12 τιμωρίων. Εμείς κρατήσαμε τις θέσεις μας. Το θέμα είναι οι πληρωμές. Η συμφωνία αυτή δυστυχώς δεν λύνει το πρόβλημα των πληρωμών, μάλιστα την χειροτερεύει. Για το 2014 πετύχαμε το ελάχιστο δυνατό. Για το 2015 έχουμε κάνει εντελώς λάθος. Δεχθήκαμε για μια ακόμη φορά να θυσιάσουμε την αναγκαιότητα των υποχρεώσεων στον βωμό των πολιτικών υποσχέσεων. Αυτά δεν είναι σοβαρά. Για του χρόνου έχουμε 145 ε, δις πληρωμές και 100, ε, υποχρεώσεις και 141 πληρωμές. Τέσσερα δις θα προσθεθούν στα χρήματα που ήδη χρηστάμε. Τα επόμενα χρόνια λοιπόν τα πράγματα θα πάνε ακόμα χειρότερα προφανώς. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε έτσι. Από αυτό θα εξαρτηθεί η αξιοπιστία της κοινότητας. Πολλά πολιτικά κόμματα μένουν στο περιθώριο ή μάλλον θέλουν να σεβαστούμε τα όρια διότι υποτίθεται λειτουργούμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι εκπρόσωποι των κομμάτων που κυβερνούν και σαν Συμβούλιο θέλουν να αφήσουν την Ευρώπη χωρίς πόρους. Η Ιταλική Προεδρία που υποτίθεται είναι υπέρ της αλλαγής και υπέρ των επενδύσεων είναι συνένοχος για μια ακόμη φορά. Τα λόγια δυστυχώς δεν ακολουθούνται από πράξεις. Για να μην πω ότι τα λόγια είναι αντίθετα από τις πράξεις. Ευχαριστώ. Η κυρία Μοντέλ δεν είναι όμως εδώ. Οπότε θα περάσω στον μεθεπόμενο που είναι ο κύριος Ρούμπεκ. 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το μικρόφωνο σας παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι ο υπολογισμός του 2015 μας φαίνει αντιμέτωπους με μεγάλες προκλήσεις. Εμείς θέλουμε από τη μια Ευρωπαϊκή Ένωση να μην υπερχρεώνεται εις βάρος των κρατών μελών ε, αλλά αυτό δεν γίνεται. Ε, τα κράτη-μέλη να μετατοπίζουν τα δικά τους χρέη στην Ευρώπη και να μην γίνεται αυτό σεβαστό στο σύμφωνο σταθερότητας. Νομίζω ότι το σχέδιο του Juncker αποτελεί μεγάλη ευκαιρία. Δηλαδή και το θέμα των ιδίων πόρων να το συζητήσουμε πιο σοβαρά κάποια στιγμή, για παράδειγμα, ε, για το φάσμα, το ραδιοφάσμα των 700 MHz, ε, να δούμε πώς θα γίνουν οι πληστηριασμοί για να δοθούν οι άδειε των συχνοτήτων αυτό και να συνδεθεί με την ε, διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη, Connecting Europe, ή με τον ε, ορίζοντα το 2020. Όλα αυτά σε ένα σύστημα SDIT είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και στις ε, ψηφιακές αγορές, τις οπτικές είναι να υπάρξει μια πραγματική ενιαία αγορά, μια ενιαία ψηφιακή αγορά και να υπάρξει και ένα κίνητρο για να εγκριθεί από το Συμβούλιο αυτό το πακέτο της ψηφιακής αγοράς. Τότε θα έχουμε προχωρήσει πραγματικά και τα νέα έργα ε, τα οποία έχουμε σκιαγραφίσει μόνο, ε, θα, αν προχωρήσουν, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις επιχειρήσεις και μεγάλο κίνητρο. Ευχαριστώ κύριε Ρούμπιχ. Πριν δώσω το λόγο στον επόμενο μιλητή μας που είναι ο κύριος Μάνκα, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι το Συμβούλιο χρειάστηκε να αποχωρήσει ε, από τη συζήτηση γιατί ε, υπάρχει μια διοργανική άλλη ανελημένη υποχρέωση, θα επιστρέψουν. απλώ ήθελα να σας ενημερώσω. Ο κύριος Μάνκα, για ένα λεπτό παρακαλώ. Συμφωνώ ε, με τον πρόεδρο της Επιτροπής, με τον κύριο Γιούγκερ, ότι πρέπει να αλλάξουμε τις ε, μεθόδους ε, εργασίας. Αυτό το μήνυμα απευθύνθηκε και στο Συμβουλίο, τουλάχιστον όσον αφορά στις δημοσιονομικές διαπραγματεύσεις. Χάρη <clears throat> στον εισηγητή, στην εισηγήτρια και στις ομάδες της, έχουμε επιτύχει συμβιβασμό. Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Από την άλλη βέβαια είναι και μια σαφής εξοικονόμηση. εξοικονόμηση προκύπτει όταν έχουμε καλύτερη δημοσιονομική πολιτική. Αυτό λοιπόν πρέπει να το συζητήσουμε περαιτέρω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και στο Συμβούλιο και με τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων. Μόνο αν εργαζόμαστε αποτελεσματικά, μόνο έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις του 21ου αιώνα, την κλιματική αλλαγή, τη φοροποφυγή, την παγκοσμιοποίηση, τις απειλές στην ασφαλεία μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενος μιλητής για 1,5 λεπτό, ο κύριος Ashworth. <clears throat> Πρόεδρε, Χαιρετίζω το γεγονός ότι αυτός ο προϋπολογισμός εντάσσεται μέσα στα συμπεφωνημένη όρια του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου. Και επίσης πολύ καλό το ότι υπάρχει μεγαλύτερη έμφαση στις ε, θέσεις απασχόλησης. Ε, κύριε Επίτροπε, δείξατε ουσιαστική πρόθεση να καλύψετε τις ανάγκες των πολιτών και σας συγχαίρω επ' αυτού. Όμως ε, απογοητεύτηκα για το ότι δεν υπήρχε καμία πρόθεση να ε, πληρωθούν οι εκκρεμούσες πληρωθούν πληρωμές. Αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι λοιπόν ε, σαφές ότι κατά το παρελθόν δαπανίσαμε και δαπανούσαμε περισσότερα από αυτά που κερδίζαμε, άρα δηλαδή οι δαπάνες ήταν μεγαλύτερες από τα έσοδα. Η απάντηση δεν είναι να ζητάμε περισσότερα έσοδα. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να χρησιμοποιούμε αποτελεσματικότερα τους πόρους που διαθέτουμε. Με πεπερασμένους πόρους πρέπει να ιεραρχούμε τις υποχρώσεις μας. Για να φτάσει όμως εκεί το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει μεγαλύτερο ρόλο ε, κατά την, τον έλεγχο κυρίως ε, του προϋπολογισμού ε, και επίσης σε μεγαλύτερο ρόλο στην αξιολόγηση της πραγματικής αξίας των πραγμάτων. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Τούρβαλτς παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ βλέπω ότι συμβαίνει εδώ κάτι το πάρα πολύ περίεργο. Ε, σήμερα θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και τους εισηγητές, όλους τους εισηγητές για την τεράστια προσπάθεια την οποία έκαναν και το λέγει αυτό ε, στις γλώσσες των εισηγητών ο κύριος Τόρβαλτς. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τους συνεργάτες μας οι οποίοι έκαναν πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Και φυσικά να ευχαριστήσω και τον πρόεδρό μας γιατί μας οδήγησε σε μια ικανοποιητική λύση. Ε, μέσα σε όλα πρέπει να πω ότι το Συμβούλιο ε, τελικά ήταν ιδιαίτερα επίμονο στην καταπολέμηση των προτάσεων ε, του του Κοινοβουλίου. Είχε ένα πείσμα σοβιετικού τύπου. Ξέρετε ότι Συμβούλιο στα ρωσικά ε, λέγεται Σοβιέτ. Ευχαριστώ για 1,5 λεπτό κύριο Σιτσενίκη. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι ευρωβουλευτές, εσείς για ποιον δουλεύετε. Αυτό δεν με απασχολεί μόνο εμένα, απασχολεί και τους πολίτες που σας έχουν ψηφίσει και πραγματικά δεν τους ρίχνω το φταίξιμο. Εδώ στο Κοινοβούλιο ε, εγκρίθηκε μια νεοφιλελεύθερη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην υπηρεσία των ισχυρών και ένας πρόεδρος που νομίζει ότι ε, ε, με φορομπηχτική πολιτική και να εκφοβίζει τον ελληνικό λαό αυτό είναι τμήμα της εντολής του. Τώρα συζητούμε για τον προπολογισμό του 2015. Είναι ένα από τα λίγα εργαλεία αναδιανομή και ε, κοινωνικής δικαιοσύνης που μας έχουν απομείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά από μια παντομήμα διαπραγματεύση, μας φαίνεται σήμερα ένα νεμικό προπολογισμό που θα συνεχίσει να καταστρέφει την ευρωπαϊκή οικονομία, να διευρύνει το φάσμα μεταξύ λαών Βορρά και Νότου και ε, δίνουν φτερά στο φάσμα του φασισμού. Αύριο το Κοινοβούλιο μπορεί να δείξει θάρρος και να απορρίψει ε, το κοντό, φθαλμό, ε, αντικοινωνικό, αντιευρωπαϊκό και προπολογισμό λιτότητας. Αύριο το Κοινοβούλιο μπορεί να διατρανώσει ότι θέλει μια Ευρώπη όπου η Ελλάδα, η Γερμανία και η Ισπανία εκτός από εμπορική εταίρη θα είναι και αδελφοί λαοί μπορεί να το κάνει αυτό ή μπορεί να συνεχίσει τον ανεύθυνο δρόμο ε, προς ε, την απαξίωση των θεσμικών οργάνων, ε, την εξαθλίωση των λαών και την παρακμή της Ευρώπης ότι εργάζεται ο Γιούνκερ για τους φορολογικούς παραδείσους, αυτό το ξέραμε. Εσείς για ποιους δουλεύετε. Αύριο θα έχετε την ευκαιρία να το αποδείξετε. Ευχαριστώ. Ε, έχει ζητήσει ερώτηση με μπλε κάρτα ο κύριος Βιώτη. Τη δέχεστε. Παρακαλώ. 30 seconds, please. Eh, Κύριε Σενίκε, κάποια από αυτά τα οποία είπατε είναι πολύ ενδιαφέροντα. Είναι ενδιαφέρουσες και οι τροπολογίες τις καταθέσατε τις τελευταίες ώρες. Είπατε ότι ήταν παντομήμα η διαπραγμάτευση. Δεν ήσασταν παρόν όμως. Γιατί θα μπορούσαμε να είχαμε ακούσει πιο σοβαρά τις απόψεις σας και από κοινού θα μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα προϋπολογισμό λιγότερο ελευθεροκτόνο όπως είπατε κι εσείς. Τι δεν κάναμε, τι έπρεπε να κάνουμε. Και θα ήθελα να σας ζητήσω αν θέλατε να πάρετε νωρίτερα μέρος. Για 30 δεύτερα να απαντήσει ο κύριος Ετσενίκη. Ήμουνα στην Επιτροπή Προπολογισμών, όπως κάθε βουλευτής, έκανα τροπολογίες εξ ονόματος της ομάδας μου και ε, η ε, εργασία της ομάδας ήταν υποδειγματική και ε, από την τοποθέτησή σας εγώ δεν δίδα καμία ερώτηση, οπότε δεν έχω τίποτα να σας απαντήσω. Thank ε, Σας ευχαριστώ για ένα λεπτό. Ο κύριος Σκέρλετς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Πάρα πολύ συχνά ε, βλέπουμε θεομηνίες και καταστροφές που πλήττουν σφοδρά ε, ορισμένες περιφέρειες της Ευρώπης με μεγάλες οικονομικές ζημίες και θύματα. Εκατομμύρια ευρώ αφιερώνονται για την καταπολέμηση των πλημμυρών. Στην Κροατία είχαμε ε, στη Σλαβωνία ε, πλημμύρες με ζημίες της τάξης των 197.000 ευρώ. Ε, καλύτερα λοιπόν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τα κονδύλια και η πολιτική συνοχή είναι η καλύτερη ε, πολιτική για να ε, μπορέσουν τα κράτη-μέλη να ανταποκρίνονται. Υποτίθεται ότι η πολιτική συνοχής προλαμβάνει την κλιματική αλλαγή, δημιουργεί και θέσεις εργασίας βιώσιμες και μπορεί βιώσιμα να βοηθάει την οικονομία μικρότερων κρατών μελών. Εδώ ε, ε, καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαδραματίσει ένα ρόλο πρωταγωνιστικό και παρακαλώ να αφοσιωθούμε όλοι σε αυτό. Κύριο Σάνοτ. Για μια ακόμη φορά έχουμε έρθει εδώ να συζητήσουμε το θέμα του προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2015. Να σας εξηγήσω πώς το βλέπουμε αυτό εμείς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχει αντίληψη ότι οι φορολογούμενοι ε, ζητείται να συνεισφέρουν όλο και περισσότερο, αλλά δυστυχώς δεν είναι ανταποδυτικά τα τέλη αυτά. Και υπάρχει και το θέμα της συνεισφοράς, της επιστροφής μάλλον, τίθεται και το θέμα της Βρετανικής συνεισφοράς ε, και δεν ξέρω σε ποιο βαθμό φαίνεται ότι η Ελλάδα και η Ιταλία πληρώνουν περισσότερα ενώ πληρώνουν λιγότερα οι Γερμανοί και οι υπόλοιπες χώρες. Το Μάιο οι τοπικές εκλογές έδωσαν ψήφους σε κόμματα οι οποίες είναι εναντίον της Ευρώπης και αυτό φαίνεται ότι είναι πλειοψηφικό στην, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μην το υποτιμάτε αυτό. Δύο δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι 58% των εκφραζόμενων απόψεων θέλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση να φύγει ή μάλλον το Ηνωμένο Βασίλειο να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, τώρα ο προϋπολογισμός είναι μια κομψή συμβιβαστική λύση ανάμεσα στο Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Είναι μια συμβιβαστική λύση την οποία πολλοί Ίσως και οι περισσότεροι από εσά δεν συμφωνούν, ακόμα και αν ίσως την δεχθούν τελικά. Ακριβώς εδώ υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα ανάμεσα σε αυτά τα οποία συμβαίνουν εδώ μέσα και σε αυτά τα οποία συμβαίνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Νομίζω ότι δεν είναι ένα συμβιβασμός τον οποίο ε, θα δεχθεί ο Βρετανικός λαός. Το χάσμα ανάμεσα στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι απλά μια λωρίδα ωραίας θάλασσας, γαλάζιας θάλασσας, αλλά είναι ε, πεπιθήσεις διαφορετικές για το τι πράγματι πρέπει να είναι η Ευρώπη. Ο κύριος Συναδεινός, ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, ένα σεισμό στη χώρα μου την Ελλάδα που προκάλεσε ζημιές περίπου 147 εκατομμυρίων ευρώ με περισσότερες από 2.500 κατοικίες να μην σε θέση να στεγάσουν αντίστοιχε οικογένειε οδήγησε την ευρωπαϊκή ένωση της αλληλεγγύης να διαθέσει περί τα τρία εκατομμύρια ευρώ ως βοήθεια. αυτή η ενέργεια αποδεικνύει το πραγματικό πρόσωπο της ευρωπαϊκής ένωσης μια ένωση που δημιουργεί κανόνες και νόμους για να τους εφαρμόζει όταν και όπου συμφέρει μια ένωση που σκέφτεται τα οικονομικά συμφέροντα των ισχυρών κρατών ενώ αφήνει τις λοιπές χώρες με ψίχουλα μια ένωση η οποία δεν μπορεί και δεν θέλει να σκεφτεί ότι μια χώρα που μαστίζεται από μια τεράστια οικονομική κρίση που η ανεργία έχει φτάσει σε απάνθρωπα ύψη και με το μισό σχεδόν πληθυσμό να ζει στα όρια της φτώχειας δεν μπορεί να αξιολογεί και να ακολουθεί τους ίδιους κανόνες με χώρες όπου δεν συντρέχουν παρόμοιες συνθήκες. είναι βαθιά και κάθετα ενάντια στην ιδρυτική διακήρυξη της ένωσης ο έκδηλος οικονομικός και πολιτικός ρατσισμός του προϋπολογισμού και το κοινωνικό έλλειμμα των κυρίαρχων δυνάμεων. ας θυμηθούμε όλοι τις αρχές πάνω στις οποίες χτίστηκε η ευρωπαϊκή ένωση την ισότητα την αμοιβαία συνεργασία και το σεβασμό. ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για μισό λεπτό ο κύριος Μούρεσαν. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, αγαπητή κυρία Επίτροπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προπολογισμό για το 2015. Δεν χωράει καμιά αμφιβολία ότι αυτό είναι ευχάριστα νέα για την Ευρώπη. Μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε ότι αν δεν είχαμε το Κοινοβούλιο θα είχαμε δημοσιονομική κρίση και ε, θα ήταν σε εμπλοκή πολλά προγράμματα εκατομμυρίων και αυτό θα ήταν αρνητικό για μικρομεσαίες επιχειρήσει, ερευνητέ και φοιτητέ. Ε, χάρη όμω στη στεναρή και ισχυρή θέση του Κοινοβουλίου καταφέραμε να ανατρέψουμε όλες τις περικοπέ σχεδόν ε, του ε, Συμβουλίου και ε, σταθεροποίησαμε τουλάχιστον τις πληρωμές όσο γινόταν, αλλά δεν έχουμε λύσει το πρόβλημα. 25 δισεκατομμύρια θα έχουν σωρευτεί στα τέλη του έτους, απλήρωτη λογαριασμοί. Χρειάζεται ένα σχέδιο για να μειωθεί, γιατί είναι απαράδεκτο. Γι' αυτό καλωσορίζω αυτή την πρόταση. Να καταρτιστεί ένα σχέδιο για να καλυφθεί αυτή η καθυστέρηση και χαίρομαι που η κυρία Γεωργίευα ε, ε, δήλωσε προθυμία να συνεργαστεί. Παραμένουν όμως και άλλα θέματα και από τα σημαντικότερα ε, αφορούν τα ειδικά μέσα. Εγώ είμαι εισηγητή για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης για τις ε, πληρωμές το 2015. Πρέπει να σας πω ότι το Συμβούλιο πιστεύει ακόμα ότι οι πληρωμέ θα πρέπει να είναι εντό των πλαισίων του προπολογισμού και για το μέσο αυτό. Άλλο ένα τρόπο με τον οποίο προσπαθεί ε, το Συμβούλιο να παρακάμψει το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Εμεί είπαμε ότι αυτά είναι έξτρα πάνω από τα περιθώρια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν επιτρέπεται να έχει ελλείμματα και να σωρεύει ελλείμματα. Θα πρέπει να εξασφαλίσει το Συμβούλιο τη δυνατότητα τη Ένωση να εξοφλεί του λογαριασμού. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, κύριο Βόν. Κύριε Επίτροπε, μιλάμε πάρα πολύ για τους ε, αριθμού για τα στοιχεία στου ε, στους προϋπολογισμούς, αλλά πολλές φορές ε, ξεχνάμε προς τι χρησιμοποιούνται τα χρήματα. Αναφέρομαι κυρίως σε όσους επωφελούνται από τις επενδύσεις, ξέρουμε ποιοι επωφελούνται από τις γεωργικές, παραδείγματος, ε, Παραδείγματο χάρη επενδύσεις, αλλά και αυτοί που εργάζονται στην Γεωργία. 750 εκατομμύρια λίρες ε, δόθηκαν στην Αγγλία ε, σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, 20 σε ένα άλλο, 40 σε ένα τρίτο. Όλα αυτά είναι προγράμματα τα οποία δεν θα μπορούσαν να εφαρμοστούν αν δεν υπήρχαν οι επενδύσεις Ευρωπαϊκής Ένωση. Άρα δηλαδή δεν είναι όλοι οι Εγγλέζοι κατά της ένωση. Βλέπουμε ότι υπάρχουν και ωφέλη. Και θα ήταν καλό ότι είναι σημαντικό όλοι μας να επενδύσουμε στην καινοτομία, στην έρευνα, στην ανάπτυξη, κυρίως στους ακαδημαϊκούς θεσμούς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον των οικονομιών μας. Για να γίνει βέβαια κάτι τέτοιο χρειαζόμαστε έναν ε, προϋπολογισμό που να είναι αποτελεσματικός και που εστιάζει στα σωστά σημεία που είναι εκείνα που προάγουν την ανάπτυξη και την απασχόληση. Για 1,5 ε, λεπτό, επόμενος ομιλητής, ο κύριος ε, Γιουζούκ. Ευχαριστώ πολύ ε, ευχαριστώ πρόεδρε. Παρά τις θέσεις του Συμβουλίου και παρά το ότι χρειάστηκε να δουλέψουμε πάρα πολύ και να προσφύγουμε και στους προϋπολογισμούς τους διορθωτικούς Το Συμβούλιο τελικά συμφώνησε στις τελικές προτάσεις του Κοινοβουλίου και στο ότι τα χρήματα από πρόστιμα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ε, στα πλαίσια των διορθωτικών προϋπολογισμών. Ε, κάτι το οποίο φτάνει περίπου τα τρία δις. αλλά από την άλλη θα έχουμε ήδη για τις πληρωμές ένα ποσό το οποίο δεν θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες μας. Ε, ε, βέβαια καταλήγουμε σε 4 εκατομμύρια, δισεκατομμύρια επιπλέον για τις πληρωμές αλλά δυστυχώς ε, το έλλειμμα είναι μεγάλο και το χρέος είναι γύρω στα 30 δις. Απαιτείται χρόνος, απαιτείται ρευστότητα και γι' αυτό με ανησυχία Άκουσα κάποιες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να χρησιμοποιηθεί το αποθεματικό γιατί όπως ξέρετε ότι το αποθεματικό αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται ε, για τομείς εκτός γεωργίας. Τι γίνεται όμως με το 2015 και τη συνέχεια του εμπάργου γεωργικών προϊόντων προς τη Ρωσία μήπως θα πρέπει να βοηθήσουμε τους γεωργούς περισσότερο από ό,τι τώρα. Ο Μαρτζή ένα λεπτό. Να ευχαριστήσω τους εισηγητές για την προσπάθειά τους. Να υπογραμμίσω την τεράστια προσπάθεια του Προέδρου Αρτουή και να σημειώσω τη συνένεση που σημειώθηκε στην Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή για να αντισταθούμε στις προτάσεις του ε, Συμβουλίου. Βέβαια ε, τα βήματα τα θετικά του Συμβουλίου είναι πάρα πολύ μικρά, ήρθαν την τελευταία στιγμή και δεν λύνουν το πρόβλημα των καθυστερημένων λογαριασμών. Γιατί το 2015 θα βρεθούμε πάντα με 26 δις ε, εκτός κάλυψης. Ήδη από τώρα λοιπόν θα πρέπει να ξεκινήσουν οι συζητήσεις με το Συμβούλιο έτσι ώστε να μπορέσουμε να βρούμε μία λύση για τα επόμενα χρόνια διότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι οι μειώσεις θα αρχίσουν να παίζουν σημαντικό ρόλο από το 18 και μετά ε, ιδιαίτερα στον τομέα της πολιτικής της συνοχής. Και αν δεν βρεθούν λύσεις από σήμερα, τότε σε λίγα χρόνια η κατάσταση θα είναι πλέον χωρίς αντιμετώπιση. Το Συμβούλιο πρέπει να βρει λοιπόν λύσεις αλλά διακόπτεται ο μιλητής από την Πρόεδρο. Ένα λεπτό. Τον λόγο έχει ο κύριος Βάλλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η συμφωνία για τον προϋπολογισμό είναι μια ήττα για όλους. Αυτό πρέπει να είναι σαφές. Και για το Κοινοβούλιο, το οποίο δεν μπόρεσε να πετύχει αυτά που ζήτησε, θυσίασε τις προτεραιότητές του, είναι μια ήττα για το Συμβούλιο και για τα κράτη-μέλη, γιατί δεν κατάλαβαν ότι τα χρέη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δικά τους χρέη. Και αυτά τα πάνω από 20 δις δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα στις επιχειρήσεις τους, στους πολίτες τους, στις διοικήσεις τους. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε σύγχυση γιατί τώρα προτείνει αριθμούς τους οποίους είχε απορρίψει κάποτε ε, είναι η κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λιτότητα από τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη ζητούν λιτότητα από την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι στριμωγμένο στη μέση και οι πολίτες είναι πολύ κουρασμένοι από όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ για 1,5 λεπτό. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Κίρτσος, παρακαλώ. Ευχαριστώ νομίζω ότι ο συμβιβασμός που επετεύχθη είναι θετικός. καταρχήν μπήκε ένα φρένο στις περισσότερες οφειλές άρα ενισχύθηκε η αξιοπιστία της ευρωπαϊκής ένωσης εξασφαλίστηκε η, χρηματοδότηση, η βασική χρηματοδότηση των πολιτικών και υπάρχει και μια εικόνα ομαλότητας γιατί θεωρώ ότι αν είχαμε, πάμε, αν είχαμε πάει σε μια κρίση προϋπολογισμού και δουλεύαμε με δωδεκατημόρια θα είχαμε ένα σωρό πρακτικά και πολιτικά προβλήματα από την άλλη πλευρά όμως ο προϋπολογισμός δεν είναι προϋπολογισμός περισσότερης ευρώπης ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. παραμένουμε σε γενικές γραμμές στο 1 του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος των κρατών μελών και δεν έχει λυθεί και το πρόβλημα των ιδίων πόρων. επομένως θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά και είναι χαρακτηριστική η επιχειρηματολογία των ευρωσκεπτικιστών και των αντιευρωπαίων οι οποίοι προσπαθούν να μειώσουν ε, τα κοινοτικά κονδύλια ακριβώς για να ενισχύσουν το επιχείρημα ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει η ευρωπαϊκή ένωση. δεν θεωρώ ότι τα λεφτά του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού είναι πεταμένα λεφτά αντίθετα είναι μια σωστή ευρωπαϊκή επένδυση σε όφελος όλων των ευρωπαϊκών λαών. ευχαριστώ. Uh, Σας ευχαριστώ για ένα λεπτό τώρα, κύριος Νεκρέσκου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους ηγητές για τις προσπάθειες που κατέβαλαν. Επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει προπολογισμό για το 2015 και καλά θα κάνει και μπράβο της. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι λύσαμε όλα μας τα προβλήματα. Ε, η συνένεση την οποία επιτύχαμε είναι και ατελής ε, υπάρχουν προβλήματα και στις πληρωμές, ανεξόφλητοι λογαριασμοί, χρέη του παρελθόντος και η προσέγγιση του Συμβουλίου στις συζητήσεις με το Κοινοβούλιο ε, ε, είναι προβληματική. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργούμε θέσεις εργασίας, να προωθούμε σχέδια, ερευνητικά προγράμματα, έχουμε ζητήματα με τους ιδίους πόρους και άλλα. Ως πάρα πολύ νέο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είμαι καταπογοητευμένος και πιστεύω ότι θα βγάλουμε τα διδάγματά μας από τη φετινή κατάσταση για τον επόμενο προϋπολογισμό. Ό,τι και να λέμε, εν πάση περιπτώσει, εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο και παρά τη θέση του Συμβουλίου και της Επιτροπής, εμείς δουλεύουμε υπέρ των Ευρωπαίων πολιτών, διότι το δικό τας ε, συμφέρον ταυτίζεται με το δικό μας. Οπότε, όταν μιλούμε για τον προϋπολογισμό, θα πρέπει πάντα με διαφάνεια να προχωρούμε. Ευχαριστώ. Ο λόγος στον κύριο Μπαρέκοφ για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Ε, κύριε Επίτροπε, από τις 19 Ιουλίου στις 2 Αυγούστου Είχαμε ε, καταστροφικές πλημμύρες ε, που κατέστρεψαν τη φτωχότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χιλιάδες Βούλγαροι παρέμειναν άστεγοι. Η κυβέρνηση Βουλγαρίας υπολογίζει τη ζημιά σε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ. Ζήτησα από τον κύριο Μπαρόζο να κάνει μια εκτίμηση και ζητήσαμε 20 εκατομμύρια ευρώ που δεν μας εδόθησαν όμως. Είπαμε λοιπόν η Βουλγαρία, η φτωχότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει πληγεί θανάσιμα ε, με θύματα πάρα πολλές οικογένειες που περιμένουν στην υποστήριξή σας. Χρειαζόμαστε χρήματα και πραγματική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι αλλιώς ε, αυτός ο προϋπολογισμός θα προκαλέσει το θάνατο ανθρώπων. Σας ευχαριστώ πολύ επόμενη ομιλήτρια για ένα λεπτό, η κυρία Μισελ. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, δεν θα πρέπει εδώ να εξοραίζουμε τα άσχημα, αυτά που δεν είναι ωραία. Τον Οκτώβριο, λοιπόν το Κοινοβούλιο τα χρήματα για το 2015, αυτά που πραγματικά μπορούν ε, να πληρωθούν, τα υπολόγισε σε 146 εκατομμύρια ευρώ και έκρινε ότι αυτά είναι απαραίτητα. Τώρα λοιπόν έχουμε 146 εκατομμύρια ευρώ που έχουν καταγραφεί στα χαρτιά. Με άλλα λόγια θα υπάρξει περικοπή στην πολιτική συνοχή, στα διαρθρωτικά ταμεία αλλά και στην παιδεία και τον πολιτισμό όπως το πρόγραμμα Erasmus Plus και Δημιουργική Ευρώπη. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι αυτό είναι ανεύθυνο και το Συμβούλιο εκ νέου μας λέει ισχύει εξής η μέθοδος. Φάε ή πέθανε κατά λέξη. Δηλαδή ή να ε, συμφωνήσουμε ή αλλιώς θα υπάρχει πραγματικό πρόβλημα. Είμαστε αναγκασμένοι να δεχτούμε έναν ε, προϋπολογισμό που δεν μας ικανοποιεί και κατά την άποψή μου αυτό για μας είναι φαρισαϊσμός. Ευχαριστούμε πολύ. Ακολουθεί ε, συνάδελφος Μαχ. Κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα προϋπολογισμό περίπου 140 δισεκατομμύρια ευρώ. Και πολλοί φιλοευρωπαϊστές λέγουν ότι είναι πολύ λίγο, λιγότερο από 1% ε, του ΕΕ των κρατών μελών. Εγώ έχω την εντύπωση ότι είναι πάρα πολλά τα χρήματα αυτά. Ε, αν ε, αποφασίζουν πολύ λίγοι άνθρωποι για 140 δις και αν δω και τι προτείνουν, πραγματικά είναι πολύ μεγάλη σπατάλη που γίνεται. Ορισμένες χώρες ε, παίρνουν λιγότερους πόρους, άλλες περισσότερες. Ε, αν δούμε ε, ποιο είναι το όφελος και το συμφέρον μας, καλό θα είναι να καταργήσουμε όλες τις εθνικές συνεισφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε ελλείμματα θα έχουν ε, οι χώρες, ούτε θα πρέπει τόσο πολύ να υπερχρεώνονται για να συγχρηματοδοτούν τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Ευχαριστώ κύριος Μαρινέσκου. Τον οποίο και δεν βλέπω. Για δύο λεπτά ο συνάδελφος Δενανό. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, στο τέλος μιας δημοσιονομικής διαδικασίας την οποία θα χαρακτήριζα χαοτική το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στριμώχτηκε ανάμεσα στην αρνητική θέση των κρατών μελών να αναλάβουν τις ευθύνες τους και σε μια επιτροπή η οποία δεχόταν συνεχώς συμβιβασμούς προς τα κάτω. Πρέπει να προεδοποιήσω την Ευρωπαϊκή Ένωση για το κίνδυνο των απλήρωτων λογαριασμών, ιδιαίτερα για τα διαρθρωτικά ταμεία εφόσον δεν προσαρμόζονται οι πιστώσεις υποχρεώσεων στο επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών, το χρέος αυξάνεται συνεχώς από χρόνο σε χρόνο. Και τελικά τίθεται να αμφισβητήσει η ιδία η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμφωνία λοιπόν για τον προϋπολογισμό του 14, 15 μάλλον, και του διορθωτικού για του 14 ήταν μεν κάτι το απαραίτητο, αλλά δεν αρκεί. Θέλω πάντως να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους εισηγητές που πάλεψαν για να καταλήξουμε στο αποτέλεσμα αυτό. Πάντως εκφράζω την ευχή να αλλάξουν τα πράγματα στο μέλλον. Οι προκάτοχοί μας εδώ ζήτησαν να υπάρχει μια αναθεώρηση του, ε, των δημοσιονομικών προοπτικών το 2016 για να δούμε ακριβώς αν μπορούν να αυξηθούν οι δημοσιονομικές δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσουμε τη μάχη για μια πραγματική ευρωπαϊκή φορολογία. Σήμερα το σύστημα του «τα θέλω όλα πίσω» δεν θα επιτρέψει να υπάρξει μια αλληλέγγυα Ευρώπη. Πρέπει με κάποιο τρόπο να βρεθούν οι ίδιοι πόροι που θα μας οδηγήσουν εκτός της κρίσης που αντιμετωπίζουμε στον προϋπολογισμό, ιδιαίτερα στις πληρωμές. Ευχαριστώ κύριε Δενανό Για ένα λεπτό Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, η δουλειά για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίρκησε πάρα πολύ. Κατορθώσαμε το συμβιβασμό αλλά δεν κατορθώσαμε τελικά να καλύψουμε το κενό στον ε, προεπλογισμό χωρίς να αυξήσουμε ε, τους, ε, τις συνεισφορές των κρατών μελών. Στον προεπλογισμό προβλέπεται αυξημένα κονδύλια για την έρευνα, την ανάπτυξη, κίνητρα για την οικονομική ανάπτυξη, θέσεις απασχόλησης και σεβασμός σε μεγαλύτερη συνοχή ανάμεσα στις περιφέρειες. Από την άλλη διερωτώ με τι θα γίνει με τις ε, κρεμούσες πληρωμές. Ε, πολλοί επιθυμούν το πρόβλημα αυτό να λυθεί από τα κράτη Μα Πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο στον τρέχοντα ε, προϋπολογισμό. 4,8 δις ε, θα δοθούν για ε, κρεμούσες πληρωμές παλαιότερων ετών. Αυτή η σώρευση των λογαριασμών και των κρεμουσών πληρωμών όμως θα παραμείνει κοντά μας. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που μιλάτε για τη Σαρδινία και για την αλληλεγγύη και στον αυτό πακέτο για το 14-15. Είναι απαραίτητη αλληλεγγύη για να υπάρξει ε, κάποια ανακούφιση ε, κυρίως από τις πλημμύρες που είχαμε στη Σαρδινία τον Νοέμβριο του 2013 και που επέφεραν άμεσες ζημιές ε, σε ύψους πάνω από 650 εκατομμύρια ευρώ. Τα 16 εκατομμύρια που προβλέπονται από το Ταμείο θα καλύψουν τις δαπάνες για την αποκατάσταση των υποδομών, το υδροελεκτρικό σύστημα. Αυτό αφορά πολλούς πολίτες που προσπαθούν να ξαναρχίσουν ζωή. Ζητώ λοιπόν και την δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ιταλικής Προεδρίας έτσι ώστε αυτά τα χρήματα να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο εκεί που χρειάζονται. Πολλές φορές οι τοπικές διοικήσεις ε, είναι αναγκασμένες να αντιμετωπίσουν τη διαφθορά κυρίως κατά τη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Άρα είναι απαραίτητο να υπάρχει έλεγχος για να διασφαλίσουμε ότι κάθε ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση της γης μας, της Ιταλίας. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μόη. Επόμενος ομιλητής, συνάδελφος Τσικού. Ευχαριστώ πρόεδρε. Όπως και η προλαλή σας, καλό είναι να θυμίσουμε ότι στον προϋπολογισμό αυτό συμπεριλαμβάνονται και τα ταμεία αλληλεγγύης που αφορούν και την δική μου περιοχή, τη Σαρδινία. Συνέβη κάτι το πάρα πολύ σοβαρό, όπως ξέρετε, με 16 νεκρούς. Υπήρξε μια τεράστια φυσική καταστροφή με τις πλημμύρες. Αύριο ελπίζω να υπάρξει μια συνεκτική ενωτική ψήφος, η οποία δεν θα αφορά μόνο την ε, Σαρδινία, αλλά και την Κροατία, τη Σλοβενία, την Ελλάδα, χώρες που έζησαν δράματα, χώρες που δημιούργησαν ακόμα πιο ε, μεγαλύτερα βάρη σε συστήματα τα οποία αντιμετωπίζουν τεράστια οικονομικά θέματα. Λοιπόν, εδώ θα πρέπει να στραφούμε προς την Ιταλική κυβέρνηση, να δούμε με ποιο τρόπο τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν σωστά. Απαιτείται διαφάνεια, αυστηρότητα και συγκεκριμένος τρόπος χρήσης. Δεν μπορούν οι πληθυσμοί αυτοί να παραμένουν σε εκκρεμότητα. Πρέπει να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους γιατί έτσι και αλλιώ έχουν πολλά προβλήματα με έκτακτες φορολογικές επιβαρύνσεις οι οποίες δεν λαμβάνουν υπόψη εξαιρέσεις για τις περιοχές που χτυπήθηκαν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βιώτη. Grazie Presidente. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στο τέλος αυτής της φάσης διαπραγμάτευσης περίπλοκης και ιδιαίτερα μακρόχρονης πρέπει να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Αρτιουή και τις συζηγήτριες και τους συζηγητές του προϋπολογισμού. Η φάση αυτή ήταν ιδιαίτερος περίπλοκη. Δεν μου αρέσει να το πω αλλά η Ιταλική Προεδρία η οποία τελικά κατάφερε να πετύχει ένα σημαντικό αποτέλεσμα κινήθηκε με πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση και αυτό θα πρέπει να το πούμε. Πάντως όπως είπα το αποτέλεσμα δεν ήταν κακό. Θα πρέπει όμως να πούμε εδώ, και αυτή είναι η αίσθηση που έχω, Υπάρχει μια κάποια μορφή έλλειψη σεβασμού απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είναι το μοναδικό άμεσα εκλεγμένο όργανο των Ευρωπαίων πολιτών. Κάτι πρέπει να γίνει ως προς αυτό. Κάποιες καθυστερήσεις, κάποιες αντιλήψεις, κάποιες συμπεριφορές ε, νομίζω τροφοδοτούν την ευρωφοβία και τον αντιευρωπαϊσμό. Το σύνολο του συστήματος μέσα στο οποίο κινούμεθα με λεπτομέρειες όπως το ότι ο προϋπολογισμός είναι πιο περιορισμένος, ότι υπάρχουν λογαριασμοί που δεν πληρώνονται, δημιουργούν ένα άσχημο κλίμα. Όταν πηγαίνουμε στις χώρες μας και μιλάμε με τους νέους, τους δήμαρχους, <clears throat> τους πανεπιστημιακούς, τους επιχειρηματίες, θα έπρεπε να είχαμε περισσότερες εγγυήσει για αυτά τα οποία λέμε, να μην δίνουμε υποσχέσεις ανεπεριεχομένου. περιεχομένου. Πρέπει να έχουμε την εγγύηση ότι τα χρέη θα πληρωθούν και οι υποχρεώσεις θα γίνουν σεβαστές. Γι' αυτό υπάρχουν ανησυχίες και για τον προϋπολογισμό που κλείνει φέτος και για τον προϋπολογισμό του 2015. Ήδη προβλέπεται για το 2015 μια συμπληρωματική επιστολή για τον προϋπολογισμό. Είναι θέματα τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη μας γιατί δεν μπορούμε να μην τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας. Ευχαριστώ πολύ για 1,5 λεπτό κύριο Κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω ρητά τις δύο εισηγήτριες. Πραγματικά ηρωικό ήταν αυτό που κατάφεραν. Και οι ερευνητές και η καινοτομία και η ανάπτυξη στην Ευρώπη θα το εκτιμήσουν. Ε, και ε, επίσης ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν ενέδωσε στη δεύτερη πρόταση για το προευλογισμό. Αλλά και στην ε, καινοτομία και αλλού ε, είμαστε σε διψήφια δισεκατομμύρια τώρα σε ανεξόφλητους λογαριασμούς. Ε, γενικοί διευθυντές και διευθυντές ε, προβληματίζονται αν επιτρέπεται να υπογράφουν καν συμβάσεις γιατί βρίσκονται στις παρυφές του δημοσιονομικού ελέγχου και των επιτραπτών. Και θέλω να πω το εξή. αυτό δεν έχει να κάνει μόνο το ενδιαφέρον μου για το Horizon Εάν το Horizon τώρα γίνει ένα λατομείο, ένα νταμάρι που θα πηγαίνει ο καθένα να κόβει λεφτά για τα νέα προγράμματα, ε, γιατί είναι πιο εύκολο ε, να λαιλατηθεί αυτό το πρόβλημα αντί να αντιμετωπίσουμε το Συμβούλιο, τότε θα έχουμε 2,7 δισεκατομμύρια που θα έχουν κόψει ε, από το 2020 ε, ορίζοντα για το πρόγραμμα Juncker. Μα αυτό είναι επιπόλαιο. Αλλάζουμε τώρα επενδύσεις, ε, αντάλλαγμα άλλε επενδύσεις. Αυτό δεν θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Ευρώπη. Χρειάζεται μια κατανομή των βαρών και να μην επιλέγεται πάντα ο απλός, ο τρόπος. Θα το πάρουμε από εκεί που τα κράτη-μέλη που δεν το διαθέτουν είναι η βάρος της καινοτομία στην Ευρώπη που θα είναι η βάση πλέον για την ανάπτυξη και για τις επενδύσεις. Ευχαριστώ κύριε Έλα. Για ένα λεπτό ο κύριος Τάγκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να δράξω την ευκαιρία για να ευχαριστήσω τους συναδέλφους ε, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήταν καταπληκτική η προσπάθεια που οδήγησε και σε λύση τελικά και ε, ε, φέτος ήταν ατέρμονες οι συζητήσεις και οι διαπληκτισμοί χρόνο με το χρόνο. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε ε, τα κράτη-μέλη, άλλα λένε και άλλα κάνουν. Διγλωσία λοιπόν των κρατών μελών είναι μια συμφωνία αυτή, αλλά λύση δεν είναι. Γι' αυτό θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο εξή, όπω έχουμε συμφωνήσει, να φέρει μια κοινή δήλωση για το πώ θα λυθεί το θέμα των απλήρωτων ε, λογαριασμών και πώ θα υπάρξει μια νέα συστηματική προσέγγιση για τον προπολογισμό για να μην έχουν αυτή τη δικλωσία τα κλάτη ε, και οι μικρομεσαίοι δεν αντέχουν. Ε, διάφορες επιχειρήσεις, άλλοι οργανισμοί περιμένουν αυτά τα χρήματα στην ε, Ολλανδία το κόμμα μου, το εργατικό κόμμα, έχει δημιουργήσει μια online ε, θηρίδα που μπορεί ο καθένας να δηλώνει τι του χρωστάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ο ε, συνάδελφος Στεχόφσκι, για μισή λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω θερμά ε, τον εισηγητή, την Επίτροπο και όλους τους άλλους που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις. Γιατί, αγαπητοί συνάδελφοι, οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι αν δεν υπάρχει σαφή σε θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι διαπραγματεύσεις αυτές θα κατέληγαν στο απόλυτο φιάσκο. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ που έχουμε μπροστά μας ε, έναν προϋπολογισμό και δεν είμαστε αναγκασμένοι να εργαζόμαστε με τα προσωρινά δωδεκαρτημόρια. Γιατί κάτι τέτοιο θα υπέσκαπτε την εμπιστοσύνη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα απειλούσε τους φοιτητές μας και τους ερευνητές μας. Και αυτό που πετύχαμε πάνω απ' όλα είναι ένα καλό πακέτο, μια δέσμη μέτρων για την ανάπτυξη και την απασχόληση που είναι πολύ καλό για το μέλλον. Σε γενικές λοιπόν γραμμές το αποτέλεσμα σίγουρα είναι ο συμβασμός Έχω βέβαια κάποιες αντιρρήσεις. Ως εισηγητή στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για τον προπολογισμό θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα θέμα που με απογοήτευσε ιδιαίτερα. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πλημμυρίδα μεταναστών από ε, εμπόλεμες περιοχές και θα αυξηθούν οι μετανάστες ε, Frontex ε, και άλλες δυνατότητες που έχουμε πρέπει να ενισχυθούν έτσι ώστε αυτοί οι θεσμοί, αυτά τα Ινστιτούτα να έχουν ε, περισσότερα χρήματα για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Γιατί ε, εφόσον θέλουμε να περικόπτουμε τα κονδύλια τότε καταλαβαίνετε ότι περιορίζονται και οι δυνατότητες μας ε, στην πολιτική ασύλου. Ευχαριστούμε πολύ. Ακολουθεί για 1,5 λεπτό στην άλφας κ. Λαμασούρ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η συμβιβαστική αυτή λύση ήταν απαραίτητη. Συγχαίρω τους πρωταγωνιστές και κυρίως τους διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου. Δεν θα μπορούσαμε να σπάσουμε την όθηση που ο πρόεδρος Γιούνκερ και το Κοινοβούλιο θέλει να δώσει στην ευρωπαϊκή πολιτική. Αλλά βυθιζόμαστε σε μια σοβαρή δημοσιονομική πολιτική. Όλα τα κράτη-μέλη και οι καλοί και οι κακοί δημοσιονομικά μαθητές συμφώνησαν για να χρηματοδοτήσουν την λιτότητά τους μέσω και του κοινοτικού προϋπολογισμού. Στην ουσία αποφάσισαν να μην βλέπουν το πρόβλημα και να το αρνηθούν. Η λύση περνάει μέσω μιας μορφής ανασχεδιασμού της χρηματοδότησης της Ένωσης. Νέοι πόροι. Εμείς υπό την Προεδρία του Μόντι προσπαθούμε να βρούμε τις σωστές προτάσεις. Δεν μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες σε επενδύσεις πρέπει να έχουμε μια δημοσιονομική δυνατότητα ίδια της ζώνης ευρώ. Ποιος θα πληρώνει και πώς. Σαν παράδειγμα θέματα όπως την εξωτερική φύλαξη, μάλλον την φύλαξη των εξωτερικών συνόρων ή την άμυνα της Ευρώπης από τον Ισλαμιστικό κίνδυνο. Καιρός είναι να δούμε τι λύσεις θα βρούμε. Ευχαριστώ πολύ. 1,5 λεπτό ο συνάδελφος Σαρβαμά arvoisa puhemies sovun saavuttaminen. πρόεδρε το να πετύχουμε συμφωνία στον προπολογισμό του επόμενου αυτό από μόνο του είναι μια ευχάριστη είδηση. Ευχαριστούμε λοιπόν όλους εκείνους ε, που ε, αξίζουν τα συγχαρητηριά μας. Είναι καλό που την τελευταία στιγμή το Συμβούλιο υπαναχώρησε και αποφύγαμε την πλήρη κατάρρευση. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι η θέση του ΕΛΚ απέδωσε. Έχουμε πλέον την διασφάλιση κοντιλίων για το πρόγραμμα Έρασμος. Έχει δοθεί προτεραιότητα ε, σε αυτά τα προγράμματα και ως εκ τούτου εγώ υποστηρίζω τα αποτελέσματα. Κατά τα άλλα δεν έχουμε και πολλά για να χαιρόμαστε διότι όλα δείχνουν ότι του χρόνου οι διαπραγματεύσεις θα είναι ακόμα πιο δύσκολες. Ε, δεν μπορεί κανείς ε, να πετύχει κάτι από το τίποτα. Ε, την τελευταία στιγμή τα κράτη-μέλη λειτουργήσαν εγωιστικά. Το εργαλείο ευελιξίας ε, και τα κατόφλια ε, δεν συζητήθηκαν, του χρόνου θα ξανασυζητηθούν. Εάν λοιπόν τα κράτη-μέλη είχαν λίγο μεγαλύτερη κατανόηση για τη σημασία των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ε, δεν θα ήταν τόσο εγωιστικά. Στη τελική ανάλυση, οποτεδήποτε εφαρμόζουμε προγράμματα με ευρωπαϊκά χρήματα, θα πρέπει να υπάρχουν μεγαλύτερε συνέργειε και μεγαλύτερη υπεραξία, γιατί κάτι τέτοιο δεν υπάρχει στη δική μα τη δημοσιονομική πολιτική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για 1,5 λεπτό η συνάδελφος κυρία Κόμη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε για τους διορθωτικούς προεπλογισμούς του 2014 και για το γενικό προεπλογισμό του 2015 αναμφισβείται ένα θετικό στοιχείο. Γιατί με τον τρόπο αυτό αποφύγαμε τα δωδεκαρτημόρια, κάτι που θα, ήταν, θα οδηγούσε σε μια πολύ περίπλοκη κατάσταση. Όμως η μεγάλη δυσκολία για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα μας οδηγεί στο να μεταρρυθμίσουμε το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι τέτοιο θα διασφάλιζε την ε, χρηματοδοτική αυτονομία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και το σύστημα θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματικό, θα μπορούσαμε να εστιάσουμε την προσοχή μα στα εφικτά αποτελέσματα αντί να δεχόμαστε τι εθνικέ επιφυλάξει. Σήμερα υπάρχουν περιορισμένα οικονομικά. Όσον αφορά το διορθωτικό του 2014 είμαι ικανοποιημένη γιατί διασφαλίσαμε του απαραίτητου πόρου. Όμω δεν συμφωνώ με την επιλογή να χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια του 2015. Η αλληλεγγύη ε, για τι ε, θεομηνίε ε, ή για την παγκοσμιοποίηση δεν θα πρέπει να έχουν όρια. Αν τα κράτη-μέλη λοιπόν ε, δεν, ε, μπορούσαν να, δεν μπορούν να βοηθήσουν θα πρέπει να παρεμβαίνει η Ευρώπη. Ένα άλλο θέμα καθοριστικής σημασίας είναι ότι η Ευρώπη πρέπει να πληρώνει τα χρέη της γιατί αν η Ευρώπη δεν δίνει το καλό παράδειγμα τότε δεν μπορούμε κι εμείς να ζητάμε από τους πολίτες να τηρούν τις προθεσμίες καταβολής των φόρων. Σε αυτή την αίθουσα έχουμε συζητήσει ε, για το θέμα της ε, οδηγίας, σχετικής οδηγίας και νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε στο θέμα που αφορά στο χρέος και ε, στα ωφέλη. Ο κύριος Πλένκοβιτς για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Αντιπρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, κυρία Γεωργίευα, Θέλω να συγχαρώ όλους τους συναδέλφους και την κυρία Ντελαβέτοβα που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις για τη συμβαστική πρόταση για τον προϋπολογισμό του 2014 αλλά και τον προϋπολογισμό του 2015. Ιδιαίτερα διότι οι διαπραγματεύσεις αυτές ε, έγιναν το δεύτερο ιδιαίτος ε, του νέου ε, πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. 145 δισεκατομμύρια ευρώ είναι η αναλήψη υποχρεώσεων. Νομίζω ότι είναι μια ισόρροπη προσέγγιση ε, σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική πειθαρχία και ε, τους στόχους που έχουμε θέσει. Νομίζω ότι θα πρέπει να δίνουμε περισσότερη προσοχή τώρα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού και στην ε, πλήρωση των υποχρεώσεων μας. Ο προπολογισμό μας ε, έχει συνδεθεί και με την κρίση φυσικά και θα πρέπει να μην παραλείψουμε την ε, σημαντική συμφωνία στο Ταμείο Λεγγύης. Ιδιαίτερα για ε, μας στην Κροατία που είχαμε μεγάλα προβλήματα με τις πλημμύρες. Πάνω από 16,5 εκατομμύρια ευρώ θα λάβει η Κροατία προς το σκοπό αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πλένκοβιτς. 1,5 λεπτό ο κύριος Βαντενκάπ. Κύριε Πρόεδρε, σήμερα πολλά ακούστηκαν. Εγώ θα ήθελα να απευθυνθώ ε, και στην Επίτροπο και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και να του συγχαρώ για τη συμφωνία για το 2015. Είναι ένα μεγάλο θετικό αυτό, ένα συν Εκεί που έχω μεγαλύτερη δυσκολία είναι οι προσαρμογές που έγιναν για το 2014. Σε τέτοιες προσαρμογές, ιδιαίτερα στο σημείο 3, βλέπω μεγάλη ένταση ανάμεσα στις πληρωμές που πρέπει να γίνουν και ε, στα ερευνητικά κέντρα μεταξύ άλλων και από την άλλη την ε, χρήση του περιθωρίου τα επόμενα χρόνια ε, και το πού θα βρούμε τα νέα χρήματα. Αυτή είναι η ένταση που σας λέω ε, ότι δεν με ικανοποιεί και τι να κάνουμε, θα πρέπει να το δεχθούμε. Στον διορθωτικό προϋπολογισμό υπαριθμών 6 για το 2014 πραγματικά έχουμε λίγο χώρο για να δούμε πώς ε, θα βελτιωθεί η επικοινωνία μας για τις υποχρεώσεις των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν γίνεται πιο δημοφιλής ε, από το γεγονός ότι ε, έχει τιμωρήσει πολλά κράτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάλιστα μέσα στο Νοέμβριο. Αυτά θα πρέπει να τα δούμε. Σας ευχαριστώ και να έχετε καλές γιορτές σας εύχομαι. Ευχαριστώ κύριε Βαντεκάπ. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Στέφανετς. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η συμφωνία για τον προϋπολογισμό του 2015 σημαίνει ότι ίσως και να πετύχουμε τους τρεις βασικούς μας στόχους, δηλαδή την κάλυψη των απλήρωτων λαγοριασμών, την χρηματοδότηση των προγραμμάτων στα κράτη-μέλη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην ανταγωνιστικότητα και στην ανάπτυξη και το περιβάλλον. Και θα πρέπει ο προϋπολογισμός να βοηθά την προσπάθεια επίτευξης αυτών των στόχων. Να μην αγνοούμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους νέους πολίτες. Ένα τομέας ο οποίος έχει αγνοηθεί λίγο είναι το θέμα της έρευνας και εδώ αναφέρομαι και στο παράδειγμα του προγράμματος Horizon. Υπάρχουν κάποια θετικά σημεία. Έχουμε 8 δις σαν παράδειγμα για την τροφοδοσία του νέου προγράμματος του επενδυτικού του κυρίου Γιούνκερ των 300 δις. Ελπίζω να βρεθούν τα περισσότερα χρήματα που απαιτούνται και αυτό να βοηθήσει λίγο και τον προϋπολογισμό. Πάντως παραμένει χαίνον το θέμα της πληρωμής ε, των λογαριασμών. Ίσως θα πρέπει να προβλέψουμε και κυρώσεις για τους απλήρωτους. Ευχαριστώ κύριε Στέφανες. Ε, ολοκληρώθηκε εδώ κατάλογος των ομιλητών. Έχουμε πολύ μεγάλη καθυστέρηση και σας παρακαλώ να τηρείτε το χρόνο που έχει συμφωνηθεί. Αυτό ισχύει και για το ΚΑΤΣΔΙ. Και πάλι έχω περισσότερες αιτήσει ε, από χρόνο ομιλία. Οπότε θα σας παρακαλέσω την κατανόησή σας, συνάδελφος Σούλιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, ε, λέει η κυρία Σούλιν, που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία. Βέβαια, εγώ δεν έμεινα ικανοποιημένη. Αντί για 7 δισεκατομμύρια επιπλέον, έχουμε μόλις 4,8 δις συμφωνήσει, ε, με τα οποία Μόλις θα σταθεροποιήσουμε τους λογαριασμούς, δεν θα τους ξοφλήσουμε. Θα πρέπει οπωσδήποτε το συντομότερο να ξοφληθούν αυτοί οι λογαριασμοί, έτσι ώστε να μπορέσουν οι δήμοι, οι κοινότητες και οι επιχειρήσεις να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Οι συμβάσεις θα πρέπει να τηρηθούν και να τιμηθούν και χωρίς οικονομικούς ε, πόρους δεν μπορεί να υπάρξει και ένα αιτήσιο προγραμματισμός για την ανάπτυξη. Ε, χαιρετίζω το σχέδιο του κυρίου Γιούνκερ για τις επενδύσεις και χαίρομαι και για το ε, Ταμείο Αλληλεγγύης που έδωσαν στην Σλοβενία 18 εκατομμύρια που θα χρησιμοποιήσουμε για την καταπολέμηση της θεομηνίας. Ευχαριστώ κυρία Σούλιν και τώρα... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Συμβούλιο μας έχει απογοητεύσει πλήρως στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό του 2015. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε μια σαφέστατη θέση και για τον προϋπολογισμό του 2014 και για το 2015. Οι υποχρεώσεις πρέπει να βασίζονται σε βεβαιότητα χρηματοδότησης. Χαίρομαι που σε κάποια σημεία που αφορούν την εξωτερική πολιτική καταφέραμε να διορθώσουμε κάπως τα πράγματα, ιδιαίτερα για την πολιτική γειτονίας και την ΚΕΠΑ. Πολιτικές πάρα πολύ σημαντικές ε, μετά τα τελευταία συμβάντα. Η μείωση τώρα του Ταμείου Εγγυήσεων στην Γεωργία είναι κάτι το οποίο θα προσθέσει προβλήματα στους γεωργούς που ήδη υποφέρουν από το ρωσικό εμπάργο. Είναι απαραίτητη η γεωργία αυτή για την Ένωση, μην το ξεχνάτε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπαλτσίτης. Ο συνάδελφος κ. Φαρία παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Ελπίζω αύριο να επιβεβαιωθεί η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε για τον προϋπολογισμό και για το 14 το διορθωτικό και για το 15 το κεντρικό. Ευχαριστώ τους συναδέλφους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που πήραν μέρος στη δύσκολη διαπραγμάτευση. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία λόγω του υψηλού επίπεδου των απλήρωτων λογαριασμών και δυστυχώς οι περισσότερες χώρες μέλη θέλουν μόνο να προκαλούν επιστροφές ε, προς τους ε, εθνικούς προϋπολογισμούς τους. Οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο κάθε χρόνο γίνονται και πιο δύσκολες. Νομίζω ότι κάποια στιγμή αναπόφευκτα θα πέσουμε στο σύστημα των προσωρινών 12 Πρέπει να πιεστούν οι κυβερνήσεις για να επενδύσουν για το μέλλον στον τομέα της ενέργειας, των μεταφορών και της καινοτομίας. Ευχαριστώ κύριο Σόλτες. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Αξιότιμα κύριε Πρόεδρε. Η απροθυμία των κρατών μελών να υιοθετήσουν τον Νοέμβριο την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον προϋπολογισμό του 2015 μας έχει οδηγήσει ως εδώ. Και ε, σχεδόν υποχρεωθήκαμε να συμφωνήσουμε για προσωρινά 12 Τα χρήματα που εξασφάλισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεν είναι αρκετά και αυτό θα έχει επιπτώσεις για όλη την Ευρώπη. Συμφωνώ με τους συναδέλφους που μίλησαν προηγουμένως, οι απλήρωτοι λογαριασμοί σωρεύονται. Έχουν τελειώσει τα έργα και δεν πληρώνονται και από το Σεπτέμβριο έχει παραλύσει το σύμπαν. Θα πρέπει και η νέα πρόταση του προπολογισμού να το αντιμετωπίσει. Δεν το λύνει πλήρω. Ξέρω ότι δεν ευθύνεται γι' αυτό η παρούσα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά κινδυνεύει να γίνει και δικό τη πρόβλημα, γιατί δεν την προβληματίζει σοβαρά το πώ θα το λύσει. Ευχαριστώ, κύριε Σόλτε. Τελευταίο, ο κύριο Μαρινέσκου στη διαδικασία του ΚΑΤΣΔΙ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ε, ζητήσω συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ήμουν σε άλλη συνεδρίαση για το νέο σχέδιο επενδύσεων. Νομίζω ε, ότι αυτό κινδυνεύει ε, λόγω του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι όλο και λιγότερο αξιόπιστος. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάθε χρόνο τα ίδια σφάλματα. Διαπραγματευτήκαμε τον προπολογισμό του 2015 ταυτόχρονα με το διορθωτικό του 2014. Παρόλο που συχνά υπογράψαμε πολλά έγγραφα που έλεγαν ότι δεν θα πέσουμε στα ίδια σφάλματα. Άλλο το Κοινοβούλιο, άλλο το Συμβούλιο. Τώρα, αν είχαμε φτάσει σε αυτά που πρότεινε το Συμβούλιο, ε, θα είχαμε πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα. Φέτος μας λείπουν 20 δισεκατομμύρια ε, και έχουμε ένα έλλειμμα, πράγμα παράνομο, το οποίο μεταφέρουμε από χρόνο σε χρόνο. Θα πρέπει του χρόνου να αποφασίσει επιτέλους για να μπει μια τάξη το Συμβούλιο, μια τάξη στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μαρινέσκο. Ολοκληρώνεται εδώ η διαδικασία ΚΑΤΣΙΑΗ και θα δώσω το λόγο στην Επίτροπο την κυρία Γεωργίευα. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ξεκινάω από τα τελευταία λόγια ότι βρισκόμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Αυτό που έχουμε δεν είναι ένας προϋπολογισμός χαράς. Ίσως να είμαστε λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, αλλά δεν έχουμε κανένα λόγο να αισθανόμαστε ότι μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες. Οι δυσκολίες εξακολουθούν να υπάρχουν. Όμως είναι ένας προϋπολογισμός ευθύνης. Ε, για όσους ε, από εσά είπατε γιατί δεν περνάμε στα προσωρινά δωδεκαρτημόρια, ας ξεχάσουμε τον προϋπολογισμό. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο πράγματα και δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Πρώτον, τα προσωρινά ε, δωδεκαρτημόρια θα μας έφερναν σε χαμηλότερο επίπεδο προϋπολογισμού απλά και μόνο διότι η βάση του 2014 είναι χαμηλότερη. Και το δεύτερο είναι ότι η πιθανότητα να εξασφαλίσουμε τα χρήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή από πρόστιμα, αυτή η πιθανότητα θα είναι πολύ μικρότερη όταν τα μπούμε στην επόμενη χρονιά. Ε, να μην ξεχνάμε την πραγματικότητα σχετικά με τον διορθωτικό υπέρ υπέρθμων 3. Τα προσωρινά δωδεκαρτημόρια όχι μόνο θα σήμαιναν μικρότερο προπληγισμό, αλλά και διότι θα είχαμε μικρότερες ενέσεις αν θέλετε που δεν θα επέτρεπαν να σταθεροποιηθούν οι απλήρωτες πληρωμές. Εγώ ανακουφίστηκα που η δύο βραχίονες ε, της ε, αρχής προϋπολογισμού μπόρεσαν να μας εξασφαλίσουν αυτό τον προϋπολογισμό που δεν είναι προϋπολογισμός χαράς αλλά είναι προϋπολογισμός ευθύνη. Και θέλω εδώ να υπογραμμίσω κλείνοντας τέσσερα σημεία. Πρώτον, ότι όσον αφορά στις, ε, στους απλήρωτους λογαριασμούς πλέον τους ελέγχουμε. Η ακρίβεια των προβλέψεών μας ισχύει. Περιμένουμε μέχρι 25 δις μέχρι το τέλος του 2014. Πρόκειται για 1,6 δις περισσότερα από αυτά που είχαμε στις αρχές αυτού του έτους. Βεβαίως θα μας άρεσε να μην υπάρχει αυτό, να έχει σταθεροποιηθεί το επίπεδο, αλλά τουλάχιστον έχουμε τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε τη χρονιά ε, χωρίς τόσες πολλές έννοιες, με για σώρευση ε, απλήρωτων λογαριασμών. Απευθύνομαι σε εσά που μιλήσατε για την ακρίβεια των στοιχείων μας. Στις διαπραγματεύσεις ε, και εδώ ε, χαίρομαι πολύ για την ομάδα μου που κάθεται από πίσω μου, μερικοί από αυτούς. Δείξαμε ότι ξέρουμε τους αριθμούς, κατανοούμε τις τάσεις και θα χρησιμοποιήσουμε τη σαφήνεια της ανάλυσης μας για να στηρίξουμε το πρόγραμμα πληρωμών έτσι ώστε αυτό να καταστεί πραγματικότητα. Τρίτον, Θέλω για άλλη μια φορά να επαναλάβω σε αυτούς που ανησυχούν για τους γεωργούς μας να τους πω ότι στη δέσμη μέτρων βρήκαμε ένα τρόπο για να μην βάλουμε χέρι, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, στην, ε, στο απόθεμα της κρίσης. Δεν το κάναμε ούτε στην περίπτωση του εμπάργου της Ρωσίας, ούτε σε περίπτωση εξελίξεων στην ε, ε, αγορά. Κάποιοι μίλησαν για το Ταμείο Αλληλεγγύης. Επειδή λοιπόν έχουμε αυτή τη συμφωνία, μπορούμε να προσφέρουμε βοήθεια στην Κροατία ε, περίπου 9 δις 9 εκατομμύρια μάλλον, στη Βουλγαρία 10,5 εκατομμύρια και στη Σερβία Επίσης θα προσφέρουμε κάποια κονδύλια γιατί αυτή τη στιγμή διεξάγονται διαπραγματεύσεις. Αυτό όμως που θέλω να σας πω είναι το εξής. Άκουσα από πολλούς από εσάς την επιθυμία τους να βελτιώσουμε την δημοσιονομική διαδικασία και του χρόνου να τα κάνουμε καλύτερα. Θα το κάνουμε αυτό. Θα δουλέψουμε καλύτερα, σκληρότερα, θα ξεκινήσουμε νωρίτερα και θα επιτύχουμε μία συμφωνία με μία πιο δομημένη ε, συμφωνία περισσότερο δομημένη. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων αυτό που με ανησύχησε είναι ότι φάνηκε ότι δεν υπάρχει η απαραίτητη εμπιστοσύνη. Για τους πολίτες μας λοιπόν, χάρη αυτών πρέπει να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη και να έχουμε πιο χαρούμενες ε, διαπραγματεύσεις ε, και καλύτερο ε, τέλος. Για άλλη μια φορά ε, σας ευχαριστούμε, Ιταλική Προεδρία, για το αίμα και υδρότα που μας προσφέρετε. Αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι ο προϋπολογισμός ευθύνης. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Επίτροπε. Ευχαριστώ πολύ που ε, εισακούσατε την έκκλησή μου γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Και τώρα εκ μέρους του Συμβουλίου έχει το λόγο ο κύριος Ντελαβέντοβα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την συζήτηση που προηγήθηκε. Ευχαριστώ και την Επίτροπο Γεωργίευα. Η επίτευξη μιας συμφωνίας για τον προϋπολογισμό του 2015 και για τους διορθωτικούς του 2014, το είπα στην αρχή, το λέω και τώρα που τη συζήτηση, δείχνει ότι πετύχαμε τους στόχους μας και ότι οι θέσεις μας δεν είναι και τόσο αποκλίνουσες. Όπως έχουμε επανειλημμένα πει, η διαδικασία του προϋπολογισμού διεξήχθη φέτος κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και μόνο χάρη στις προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων καταφέραμε να βρούμε μία λύση για ένα ρεαλιστικό και ισόρροπο προϋπολογισμό για το επόμενο έτος. Ταυτόχρονα μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε και το θέμα των απλήρωτων λογαριασμών. Η Ιταλική Προεδρία είναι ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα στο οποίο καταλήξαμε και σας ευχαριστώ όλους για το πνεύμα ε, το συμβιβαστικό το οποίο επιδείξατε. Βέβαια συνειδητοποιούμε, όπως άλλωστε περιλαμβάνεται και στις κοινέ δηλώσεις για την υιοθέτηση του προϋπολογισμού, ότι έχουμε πάρα πολλή δουλειά για το 2015 και ελπίζω τη δουλειά αυτή να την ολοκληρώσουμε με το ίδιο επικοδομητικό πνεύμα που χαρακτήρισε την τελική φάση των τελευταίων διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντελαβέντοβα. Και τώρα ξανά οι συγητές, δύο λεπτά. Εκαστός αρχίζει η κυρία Γκαρδιασάβα Ρουβιά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η συζήτηση που είχαμε είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και κατέδειξε σαφέστατα τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου όλο αυτό το χρόνο που ε, εργαζόμαστε για τον προπολογισμό, ιδιαίτερα ε, στις διαπραγματεύσεις που είχαμε και με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής. Όλοι οι ομιλητές αναφέρθηκαν στο οξύτατο πρόβλημα που έχουμε με τους απλήρωτους λογαριασμούς. Άλλοι είμαστε πιο φιλοευρωπαϊστές και πιο ενθουσιώδεις, άλλοι λιγότερο. Αλλά όλοι όσοι μιλήσαμε αναφέραμε το σοβαρότατο πρόβλημα που υπάρχει με τους του λογαριασμούς. Από την 1η Πρώτου λοιπόν το 2015 θα πρέπει να αρχίσουμε να εκπονούμε αυτό το σχέδιο στο οποίο έχουμε αναποθέσει τόσες ελπίδες και στο οποίο τόσο πολύ πιστέψαμε για να συμφωνήσουμε που σας είπα δεν είναι ικανοποιητική αυτή η συμφωνία, τουλάχιστον για το Κοινοβούλιο. Γιατί εμείς πιστεύουμε ειλικρινά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα και με καλύτερο προπολογισμό. Και εγώ επειδή είμαι Ευρωπαίστρια και πιστεύω ότι ο Ευρωπαϊκός προπολογισμό μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ το ευρωπαϊκό εγχείρημα, γι' αυτό δεν έχουμε ικανοποιημένοι με τη συμφωνία που επιτύχαμε. Αλλά και χωρί συμφωνία δεν θα είχαμε και προπολογισμό. Ούτε ανθρωπιστική βοήθεια θα είχαμε, ούτε υποτροφίε εράσμου και όπω είπε και ούτε καν χρήματα για να πληρώσουμε ε, την ενίσχυση για τους 6.000 ανέργους που σήμερα το πρωί ψηφίσαμε και θα πρέπει να είμαστε και συνεπείς εκεί. Άρα, απομένει πάρα πολλή δουλειά. Το 2015 θα είναι κρίσιμη χρονιά. Γιατί? Αν καταφέρουμε να έχουμε ένα σχέδιο που ουσιαστικά να λύνει αυτό το ζήτημα των απλήρωτων λογαριασμών, μπορούμε να πούμε στα επόμενα χρόνια σε άλλες διαπραγματεύσεις από καλύτερη αφετηρία. Γιατί το χειρότερο δεν ήταν οι αριθμοί, το χειρότερο στις διαπραγματεύσει ήταν η στάση του Συμβουλίου. Είδαμε πως δεν μπορούσε να καταλήξει σε διαπραγματευτική γραμμή. Είδαμε ότι κάποιες χώρες ανησυχούσαν περισσότερο για το πώς θα πάρουν τα λεφτά τους πίσω παρά πώς θα λύσουν τα προβλήματα της διπλανής τους χώρας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία ε, Γκαρδία Σάμπαλ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Χόλμαγερ για δύο λεπτά. Κομισάριν, liebe Ratspräsidentschaft, liebe Kolleginnen und Kollegen. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να πω ένα θερμό ευχαριστώ ε, για αυτή την δύσκολη, πετυχημένη όμως δουλειά και θα ήθελα να αναφερθώ ε, κυρίως σε αυτά που είπε στην Άρφος Άιντερ, δηλαδή ε, στο μέλλον στην Ευρώπη θα μας ρωτούν κατά πόσον είμαστε πρόθυμοι να επενδύσουμε σε έρευνα και ανάπτυξη και δεν θα μας ρωτάνε για παλιούς λογαριασμούς, άρα δηλαδή πρέπει να λύσουμε και τα δύο προβλήματα και τον, ε, την εξόφληση των απλήρωτων λογαριασμών αφενός, αλλά ε, και ε, την, την επιτυχή, τον επιτυχή, την επιτυχή διαχείριση των πόρων. Το πακέτο για την καινοτομία δεν θα πρέπει ε, να είναι εις βάρος άλλων ε, τομέων, αλλά να χρησιμοποιήσουμε κονδύλια από άλλους τομείς και αυτό πρέπει να το συζητήσουμε στο μέλλον, γιατί για μένα αυτό που έχει σημασία είναι στην Ευρώπη, στον τομέα της πληροφορικής, ε, των τεχνολογιών του μέλλοντος, στον τομέα της πληροφορικής, στον τομέα της αεροπλοείας ή της ανεξαρτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα ανταγωνισμού σε οποιοδήποτε εν πάση περιπτώσει τομέα πρέπει να προβληθούμε. Αλλιώς ε, θα ενισχυθεί περαιτέρω ο ανταγωνισμός. Πρέπει να προγραμματίσουμε προσεκτικά τον προπλογισμό. Έχει γίνει ένα βήμα, πρέπει να ακολουθήσουν και άλλα. Κατόπιν τούτου ευχαριστούμε θερμά, αλλά το ξέρουν όλοι και το ξέρουμε κι εμείς, ότι ακόμα υπολείπονται πάρα πολλά. Ευχαριστούμε την κυρία Χολμάιερ. Ακολουθεί ο συνάδελφος κυρίως Ντεπρέ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητέ Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι, αύριο θα γυρίσουμε σελίδα, τουλάχιστον για το 2014 και το 2015. Δεν έχει νόημα τώρα να μετανιώνουμε. Τι να μετανιώσει αυτό, δεν είναι, η μεταμέλεια δεν είναι στη πολιτική. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να στραφούμε προς το μέλλον και να ασχοληθούμε με αυτό. Και νομίζω ότι υπάρχουν τα εξή ζητήματα σημαντικά για το μέλλον. Πρώτο, για το άμεσο μέλλον. Επιτύχα μια συμφωνία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων για να εξοφληθεί ε, αυτό το θέμα, να καλύψουμε τους απλήρωτους λογαριασμούς, να δημιουργηθεί αυτό το σχέδιο να γίνει πραγματικότητα και όλα τα θεσμικά όργανα να σεβαστούν τις δεσμεύσεις τους. Δεύτερον, για πιο μεσοπρόθεσμα, το είπαν πολλοί ομιλητέ, μα είναι προφανές, το σημερινό σύστημα σιγά, σιγά φτάνει σε παράλυση και θα καταλήξει σε αδιέξοδο αυτό το σύστημα που βασίζεται στις εθνικές συνεισφορές. Άρα, για τους ίδιους πόρους, τι θα γίνει, ε, ε, θα γίνει πολιτική έκτακτη ανάγκη αυτό, επίγον θέμα. Τα κράτη-μέλη θα γίνουν και οι ηγέτες τους μικρές Μάργαρετ Θάτσερ που θα ζητάνε τα λεφτά τους πίσω και σιγά σιγά θα ε, σε τείχο. Και ποιο μακροπρόθεσμα ανησυχώ. Εγώ είμαι πεπισμένο ότι η υποστήριξη των πολιτών για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό δεν πρόκειται να αυξηθεί αν συνεχίσουμε στην ίδια λογική. Ούτε οι βασικέ πληρωμέ περνάνε από ενδιάμεσου φορεί που ξεχνούν να πούν στου πολίτε ότι αυτά τα λεφτά τα παίρνουν από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Είμαι πεπισμένο ότι αν θέλουμε ε, ενώπιον στην κοινή γνώμη να ε, νομιμοποιήσουμε περισσότερο τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό θα πρέπει να υπάρξει μια άμεση σύνδεση με τον Ευρωπαίο πολίτη. Δεν είναι του παρόντος αλλά θα πρέπει να καταλαβαίνει ότι τα λεφτά έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς όφελος όλων από μια κοινή προσπάθεια. Εν πάση περιπτώσει ευχαριστώ την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ήταν μεγάλη εμπειρία ε, ε, και είμαι πολύ περήφανος που συνεργάστηκα με τις δύο εισηγήτριες που ευχαρίστησα και προηγουμένως. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ντεπρέ. Για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση αυτή, ο κύριος Λεβαντόφσκι. Αυτά τα οποία συμφωνήθηκαν για το 2014 και το 2015 είναι ένας χαρακτηριστικός συμβιβασμός. Κανένας δεν είναι ικανοποιημένος. Αναβλήθηκε η συζήτηση στα σοβαρά προβλήματα, υπήρξε μια σταθεροποίηση σε κάποια θέματα δημοσιονομικά. Ε, θα ανησυχώ για το πρόγραμμα αποπληρωμής των χρεών γιατί θα πρέπει να δούμε ακριβώς πώς θα κατανοήσουν την κατάσταση η οποία γίνεται δραματική τα κράτη-μέλη. Για τους ιδίους πόρους απαιτείται μεγαλύτερη διαφάνεια, απαιτούνται περισσότερες γνώσεις και να δούμε και ποιο είναι και το κόστος της καθυστέρησης. Ε, ο σιδηρούς κανόν μέχρι τώρα είναι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός μέχρι την 1η Δεκεμβρίου να έχει πληρώσει τα πάντα. Τώρα όμως δυστυχώς αποκλίνουμε από τον ε, κανόνα αυτό. Δεν είναι καλό αυτό. Ελπίζω τον επόμενο χρόνο ε, θα είναι η κατάσταση καλύτερη, θα ειναι η κατασταση καλυτερη θα παρακολουθησουμε προσοχή το τι θα γίνει. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση αυτή. Η κοινή αύριο θα γίνει ψηφοφορία. Επόμενο θέμα σήμερα σε διάταξη. Δηλώσει του Συμβουλίου και τη Επιτροπή με θέμα την ανεπάρκεια πόρων για το σχέδιο χορήγηση βοήθεια του Παγκόσμιου Επιστημικού Προγράμματο προ του Σύρου Πρόσφυγε. Ο κύριο Ντελαβέντοβα, πρώτο εξ του Συμβουλίου. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε.